Καλημέρα σας. Μπορείτε να καθίσετε, σας παρακαλώ. Νομίζω ότι καθότι έχουμε ήδη καθυστερήσει Καλό θα ήταν ε, να πάρουμε την ε, ε, μπορούμε να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο διότι έχουμε την ψηφοφορία μόνο την Τρίτη και θέλω εδώ να ευχαριστήσω τον, ε, ε, την ε, κυρία η οποία έχει επιλεγεί σαν υποψήφιος για τη θέση εκτελεστικού διευθυντού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χρήματα Αγοράς. Καταρχήν μπορεί να μας κάνει μία παρουσίαση, μετά θα έχω με τις ερωτήσεις από τις πολιτικές ομάδες και ένα λεπτό για ερωτήσεις και στη συνέχεια η Βερένα θα έχει χρόνο για να απαντήσει των προτέρων. Ε, έχω μία ερώτηση και συμφώνησα με τον Ζων Πολ ότι θα μπορέσει να κάνει δύο ερωτήσεις, μία εισαγωγική και μετά ε, δηλαδή αντί να κάνει μία στην αρχή και μία στη συνέχεια ε, θα έχει ε, δύο διπλό χρόνο για να κάνει δύο ερωτήσεις μαζί και η Βερένα θα, θα έχει επίσης διπλό χρόνο για να το απαντήσει αν το χρειαστεί. Έχετε τα βιογραφικά και χωρίς περαιτέρω σχόλια δίνω το λόγο στην Βερίνα, Βερένα Ρώσου. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ε, βουλευτές, καλημέρα σας. Σήμερα το πρωί αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή για να μιλήσω για τις δυνατότητες να αναλάβω τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της ΕΣΜΑ. Καταρχήν θα σας μιλήσω γερμανικά που είναι η μητρική μου γλώσσα για να σας πω λίγα λόγια σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χρηματοοικονομική Εποπτεία και πώς νομίζω ότι μπορώ να συμβάλλω. Μετά θα μιλήσω αγγλικά και θα κάνω μία σύντομη περιοχή περιγραφή των καθηκόντων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει κατά τη γνώμη μου η ΕΣΜΑ. Καταρχήν η δημιουργία αυτών των, οργανισμών σημαίνει μεγάλη πρόοδο όχι μόνο για τις χρηματαγορές αλλά και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και τους επενδυτές. Διότι η κρίση μας απέδειξε ότι η χρηματοοικονομική μας εποπτεία σε γενικές γραμμές πρέπει να βελτιωθεί και όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε η ΕΣΜΑ με τα διάφορα ε, έργα της και ναι μεν μπορούμε να βελτιώσουμε την εργασία που έχει ήδη ξεκινήσει η ΣΥΖΑ αλλά επιπλέον θα πρέπει αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή με τις ευρωπαϊκές της αρμοδιότητες να αναζωογονηθεί και καταρχήν ε, αυτό οφείλεται σε μεγάλο μέρος σε εσάς. Έχουμε πολλές προσδοκίες και για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτές τις προσδοκίες πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ουσιαστικά πέντε στοιχεία οικοδόμησης. Να έχουμε μία έμπειρη και καλή ομάδα διοίκησης που θα μπορέσει να βελτιώσει και να προωθήσει αυτή την οργάνωση σε πραγματική ευρωπαϊκή εποπτεία. Δεύτερον, την καθημερινή πείρα για την εποπτεία των διαφόρων εμπλεκομένων στις χρηματαγορές επικαθημερινής βάσεως τρίτον χρειάζονται οι δυνατότητες για να υπάρχει ενιαίο έργο και το, να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε και να το εκτελέσουμε και χρειαζόμαστε ε, συ, ε, ορισμένους μεσολαβητές για να μπορέσουν να μας συνδέσουν με τις εθνικές αγορές και να εφαρμόσουν τα, τα διάφορα προγράμματα και επιτέλους θα χρειαστούμε γρήγορη αντίδραση για να εφαρμόζουμε τα προγράμματα και να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές. Νομίζω ότι μπορείτε να δείτε ότι έχω αυτές τις δυνατότητες και μπορώ να τις εφαρμόσω γιατί ε, είμαι Γερμανίδα, έχω εργαστεί επί πολλά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο και για μένα όνειρό μου θα είναι να δω να αναπτύσσεται ο οργανισμός τον οποίο ήθελα να προωθήσω. Τώρα μπορώ να σας ε, ε, να συνεχίσω αγγλικά σχετικά με τις εμπειρίε της ΕΣΜΑ για να είμαστε βέβαιοι ότι όντως θα υπάρχει μια σωστή εποπτική εργασία και καθημερινή δραστηριότητα προς τις διάφορες, ε, τους διάφορους οργανισμούς βαθμολόγησης διότι θα έχουμε άμεσες εποπτικές ευθύνες. Δεύτερον, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ε, σύνολο κανόνων το οποίο θα εφαρμοστούν κατά τρόπον ώστε να μην ε, υπάρχει ε, το αρμπιτράζ και να μην υπάρχει η διαφορετική αντιμετώπιση των διαδικασιών σε κάθε χώρα κατά τρόπον ώστε να προστατεύσουμε πραγματικά τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Τρίτον, πρέπει να βελτιώσουμε την προστασία του καταναλωτή καταναλωτή όχι για να έχουμε περισσότερη εκπαίδευση ε, των ε, καταναλωτών που ασχολούνται με τα χρηματοοικονομικά αλλά για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις ε, εξουσίες που έχουν ανατεθεί στην ΕΣΜΑ για να μπορέσει να αποκλείσει ορισμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα ή διαδικασίες. Τρίτον, με τις εποπτικές αρχές και την Ευρωπαϊκή τράπεζα ε, επενδύσεων θα πρέπει ε, να προχωρήσουμε και να είμαστε βέβαιοι ότι θα συνδυάσουμε ε, σε όλα τα επίπεδα την εφαρμογή των κανονισμών για να υπάρχει μια συνέπεια και συνέχεια εις τις πράξεις μας αλλά και στην παρακολούθηση του ρυθμιστικού συστήματος και επιπλέον θα πρέπει να ε, μπορέσουμε να προσφέρουμε μία προστιθέμενη αξία διότι θα πρέπει και να είμαστε υπόλογοι και υπεύθυνοι και θα είμαστε υπόλογοι έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πράγμα το οποίο είναι κάτι πολύ βασικό και γι' αυτό θέλω να συνεργαστούμε και να έχουμε έναν αποτελεσματικό διάλογο τον οποίο ελπίζω ότι θα ξεκινήσουμε σήμερα και προσβλέπω στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όπως σας είπα, τον λόγο έχει καταρχήν ο Ζων Πολ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Ρος, καλώς ήρθατε στην ε, Επιτροπή μας. Σε καμία περίπτωση δεν αμφιβάλλω για τις ικανότητές σας. Θα ήθελα απλώ να επενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε πολύ σημαντικές μάχες εναντίον συγκεκριμένων κρατών μελών προκειμένου να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας. Δεν καταφέραμε να πετύχουμε όλα τα οποία θέλαμε να πετύχουμε, έτσι λειτουργεί άλλωστε ο συμβασμός. Θέλουμε όμως να υπάρχουν συγκεκριμένες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει με την ΕΣΜΑ. Η ΕΣΜΑ έχει άμεσες αρμοδιότητες εποπτείας όσον αφορά τους οίκους βαθμολόγησης αξιολόγηση. Το 2009 κατάφερα να το πετύχω εγώ με την υποστήριξη των συναδέλφων μου και επίση η ΕΣΜΑ θα δραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο για την IMF και επίσης θα πετύχει ένα πολύ, πολύ σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά τα clearing houses. Ήταν πολύ ωραία αυτά τα οποία είπατε, ακούστηκαν πολύ ευχάριστα. Το πραγματικό μου ερώτημα τώρα είναι τι ρόλο θα δραματίσετε εσείς στα πλαίσια της ΕΣΜΑ ήσασταν ε, για 10 χρόνια εργαζόσασταν στην FSA, στην ε, Αρχή Εποπτείας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, στα πλαίσια της οποίας η προσέγγιση η οποία ακολουθήθηκε δεν ήταν ευρωπαϊκή. Θα μπορούσατε να εργαστείτε εσείς προς το στόχο αυτό, προς ένα ευρωπαϊκό στόχο χρησιμοποιώντας τις δικές σας αρμοδιότητες και σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν είναι φιλικό προς μια ευρωπαϊκή εποπτεία, προς μια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή, πολύ φοβάμαι ότι δεχομένως να μην έχετε εσείς την απαραίτητη εξουσία, πυγμή, δεν λέω ότι δεν θα έχετε τις ικανότητες, μπορεί να μην έχετε όμως την απαραίτητη εξουσία προκειμένου η ΕΣΜΑ να καλύψει όλες τις αρμοδιότητες τις οποίες πρέπει να καλύψει και τις οποίες άλλωστε προβλέπει ο νομοθέτης. Έχετε εσείς το κύρος αυτό προκειμένου να αντιταχθείτε στις αμφιβολίες μου αυτές, να τις διαψεύσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκοζές. Νομίζω ότι μπορώ να σας απαντήσω γερμανικά εάν ε, συμφωνείτε. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι η αρχή της ΕΣΜΑ και το κύρος της θα πρέπει να επιβληθούν ευθύς εξ αρχής γιατί θα πρέπει να διεκπεραιώνουμε επί ευρωπαϊκής βάσεως τις διάφορες ενέργειές μας και γι' αυτό θα εγώ εργαζόμενη για την ΕΣΜΑ θα είμαι ε, υπάλληλό τη, δεν θα έχω να κάνω τίποτα πλέον με την τωρινή οργάνωση όπου απασχολούμε και θα είμαι υπέρ της Ευρώπης και θέλω να προωθήσω την ευρωπαϊκή εποπτεία. Είπατε ε, ε, εν συντομία, αναφερθήκατε μάλλον στο ε, έγγραφο της FSA, είναι ένα έγγραφο αυτού του οργανισμού, όχι δικό μου και έχει δημιουργηθεί με, ως απάβγασμα των διαφόρων απόψεων που εκφράζονται στην FSA. Εγώ έχω συνεργαστεί για λογαριασμό της FSA με την Επιτροπή Λαμφαλούση και με τους εθνικούς σχετικούς οργανισμούς πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι όντως στηρίζω την προσπάθεια να επιτύχει κάτι η Ευρωπαϊκή Αρχή. Όταν θέλετε να σας πω πώς θα προωθήσω την αρχή αυτή θα ήθελα να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι ιδίω σκέφτομαι ότι αν είμαι εκτελεστική διευθύντρια θα χρειαστώ ένα προσωπικό και ε, ένα όραμα που θα πρέπει να ε, διέπουν τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργαζόμαστε με τις εθνικές αρχές αλλά και θα αντιμετωπίζουμε τις αρχές αυτές. Θα πρέπει πραγματικά να είμαστε Ευρωπαίοι και να έχουμε μια ευρωπαϊκή εποπτεία. Και αυτό νομίζω ότι καταρχήν ε, ε, πρέπει να καθοριστεί ε, με το όραμά μας με τον Στίβ Μάγιορο σαν εκτελεστικό διευθυντή και με μένα εάν με προσλάβετε και εσείς σαν κοινοβούλιο έχετε διάφορες δυνατότητες να καθορίσετε το έργο της ΕΣΜΑ και το έχετε ήδη πράξει δηλαδή πώς θα αντιμετωπίζει τους εθνικούς ρυθμιστές και νομοθέτες, πώς ε, θα ε, ρυθμίζουμε ε, και θα διευκρινίζουμε τα σημεία που είναι ασαφή μεταξύ εθνικών αρχών και Ευρωπαϊκής Αρχής, πώς επιπλέον θα γίνεται η εποπτεία των οργανώσεων βαθμολόγησης και των credit των ε, Credit Trading Organizations για να μπορέσει να υπάρξει όντως μια διαμόρφωση ευρωπαϊκής γνώμης. Ευχαριστούμε πολύ. ήταν πολύ ε, σύντομοι στην απάντησή σας. Κερδίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο χρόνο. Η επόμενη ερώτηση είναι από την Ελίζα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά σας έχουμε εδώ μαζί μας κυρία Βερένα Ρώσο. Είστε γυναίκα, ξέρουμε βέβαια ότι δεν σας επιλέξαμε επειδή είστε γυναίκα, αλλά επειδή είστε πάρα πολύ ικανοί. Πάντως η γυναική αυτή διάσταση είναι κάτι το θετικό. Οι ερωτήσει που έχω να κάνουν είναι οι ακόλουθες. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση συνέχεια τα όσο είπε ο κύριος Γκοζές. Διακυβεύονται πολύ σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στις αγορές για τις οποίες μιλάμε. Πώς εσείς θα καταφέρετε πραγματικά να προωθήσετε μια ευρωπαϊκή διάσταση. Πώς θα καταφέρετε να πετύχετε μια ευρωπαϊκή συνένεση εφόσον κάθε ρυθμιστική αρχή θα έχει τη δυνατότητα να θέσει βέτο. Πώς θα καταφέρετε εσείς να συγκεράσετε τις διαφορετικές ενδεχομένω τάσει. Δεύτερον, για πρώτη φορά πρέπει να καθορίσουμε μία εποπτεία σε κοινοτικό επίπεδο. Για παράδειγμα, για την IMF, αλλά καθώς επίσης και για τα credit ε, rating agencies, θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή εποπτεία. Πώς θα μπορέσετε εσείς να ρυθμίσετε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις αρχές αυτές. Η οίκη αξιολόγησης και για τα IMF. Πώς θα καταφέρετε εσείς να ρυθμίσετε τις αρχές αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, on Σχετικά ε, μπορώ να ξεκινήσω με τις τελευταίες ερωτήσεις και μετά μπορείτε να επανέλθετε αν δεν έχω απαντήσει σε όλα. Καταρχήν, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό η ΕΣΜΑ να επανδρωθεί με προσωπικό που θα καταλαβαίνουν καλά πώς λειτουργούν οι διάφορες αγορές στην Ευρώπη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους με τους οποίους να καταρτήσουμε κατευθυντήριες γραμμές και να διατυπώσουμε μία νομοθεσία η οποία θα ανταποκρίνεται στις διάφορες, διαφορετικές ανάγκες των διαφόρων αγορών. Επίσης δεν θα πρέπει να είναι μία συγκέντρωση από συμφωνίες στον κατώτατο παρανομαστή που θα διέπει το σύστημα αλλά είναι πολύ σημαντικό η ΕΣΜΑ να έχει όντως τη δυνατότητα να αναβαθμίσει το ρόλο της και να δημιουργήσει ε, ρυθμιστικά, ρυθμιστικές προδιαγραφές και κανονισμούς που θα είναι εξέχοντες και θα μπορούν να συγκριθούν και διεθνώς με το σύστημα το οποίο υπάρχει και να μπορέσει όντως να, όπως είπατε να ε, αναφερθεί ή στις, οργανισμού στις ε, οργανισμούς πιστοληπτικής βαθμολόγησης της ικανότητος και να ε, εξασφαλίζει ότι και οι κυβερνήσεις καλύπτουν τις ε, προδιαγραφές σε όλους τους τομείς για να μην έχετε προβλήματα στην ε, καθημερινή εποπτεία διότι ξεκινήσατε επί βάσης. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει μία αυστηρή εποπτεία, θα πρέπει όντως να ε, αμφισβητείτε τη διοίκηση και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και όσον αφορά το θέμα των διακανονισμών ξέρω ότι είναι δύσκολο διότι δεν χρειάζεται μόνο να γνωρίζετε τη δουλειά αλλά να μπορέσετε να λαμβάνετε και ψύχρεμες σωστές αποφάσεις και να επιμείνετε στη θέση σας. Ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτηση είναι η Σιλβί Γκουλάρ. Με συγχωρείτε, έχω χρησιμοποιήσει αντίστροφα το έγγραφό μου. Καλημέρα σας κυρία Ρος. Τι ωραία Σήμερα όχι μόνο μιλάμε γερμανικά, αλλά μιλά γερμανικά μια κυρία. Δηλαδή ούτε χριστουγεννιάτικο δώρο να ήταν αυτό για όλους μας. Θα συνεχίσω γερμανικά, δεν έχω τίποτα εναντίον σας και πέρσι όταν ήμουν εισηγήτρια για το ESRB συναντηθήκαμε στο Λονδίνο και γνωρίζω ότι είσαστε μια ικανότατη γυναίκα όσον αφορά τις επαγγελματικές σας Έχω όμως μια ανησυχία. πρέπει οπωσδήποτε και είναι ευθύνη μας να εξασφαλίσουμε ότι δεν διαχειριζόμαστε την κρίση αυτή σαν να είναι μια καθημερινότητα κάτι συνηθισμένο. Στα γαλλικά λένε ότι οι ε, λαθροκυνηγοί είναι οι καλύτεροι δασοφύλακες. Δηλαδή, αυτός ο οργανισμός, δηλαδή αυτός ο οργανισμός για τον οποίο μιλάμε, που ε, θεωρήθηκε στο παρελθόν από την ομάδα Ντελαροζιέ ως ένας από τους βασικούς οργανισμούς που οδήγησε υπέτειος αυτής της κρίσης τώρα με, ευρωπαϊκό, με ευρωπαϊκή σύσταση πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω από εσά συγκεκριμένα ποια είναι η πρώτη σας προτεραιότητα. Τι θα πράξετε ως προτεραιότητα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια καινούργια φάση δραστηριοτήτων. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρος, ε, αυτό το οποίο εγώ προσωπικά έμασα από αυτή την κρίση και τα τελευταία χρόνια, τέσσερα-πέντε χρόνια, είναι ότι κάναμε πάρα πολλά λάθη. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι. Ε, ε, όλοι κάναμε λάθη και ε, νομίζω είναι και σωστό, είναι έντιμο να το παραδεχτούμε δημόσια. Έμαθα όμως πολλά. Τα παθήματα μαθήματα όπως λέμε και έμαθα κυρίως ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στη διαχείριση των ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοοικονομικών φορέων. Πρέπει να επαγρυπνούμε συνεχώς και να εξασφαλίζουμε ε, το, το, σεβασμό των κανονισμών και όλων των συναφών διατάξεων από αυτούς τους οργανισμούς, τις αρχές και τους φορείς πρέπει να εξασφαλίσουμε μια σταθερότητα στις αγορές, στις χρηματαγορές και προς όφελος των πολιτών αλλά και των επενδυτών. Ήδη ε, ανέφερα ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες για τις χρηματαγορές και ε, η ΕΣΜΑ έχει ακριβώς αυτή την ευθύνη. Τη συλλογή, διαχείριση, ανάλυση και ε, ε, χρήση αυτών των αξιόπιστων ε, στοιχείων, δεδομένων που προέρχονται από τις χρηματαγορές. Λοιπόν, συλλογή στοιχείων, δεδομένων. Δεύτερον, πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίσουμε την συνετή και σωστή εφαρμογή των οδηγιών. Αυτό που πιστεύω δημιουργεί ένα πρόβλημα είναι ότι είχαμε υπερβολικές ε, ρυθμιστικές διατάξεις, ε, πάρα πολλές σωρία ρυθμιστικών διατάξεων και τις οποίες χρησιμοποιούσαμε επιλεκτικά και εν μέρη. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό το δάσος των ρυθμιστικών διατάξεων για να μπορέσουμε συνεπώς να εφαρμόζουμε την οδηγία και όλες τις ε, διατάξεις αυτές οι οποίες θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε την κρίση. Λοιπόν, συλλογή στοιχείων και σωστή εφαρμογή των διατάξεων και οδηγιών. Ευχαριστώ. Ο, ε, η κυρία Βίμπερν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι αγορές είναι παγκόσμιες και βεβαίως υπάρχει πρόβλημα ρευστότητα σήμερα που καταδεικνύει ότι οι διεθνείς εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συνεργάζονται στενά όχι μόνο σε περιόδους κρίσεων αλλά και ιδίως σε περιόδους όπου δημιουργούνται ε, νέα νομοθετικά πλαίσια για τις ε, μελλοντικές ε, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Μπορείτε να μας πείτε εσείς, αν γίνετε διευθύντρια τη ΕΣΜΑ, πώς θα αναπτύξετε και θα στηρίξετε περαιτέρω την παγκόσμια διάσταση και δεν θα ξεχαστεί. Ευχαριστώ κυρία Ρος. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό, όπως ήδη ανέφερα, να ενδυναμώσουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής Διεθνώς ξέρουμε ότι οι χρηματαγορές ε, πλέον δεν είναι μόνο ευρωπαϊκές αλλά και δεν δραστηριοποιούνται μόνο στην ευρωπαϊκή επικράτεια αλλά ε, σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό ε, θα πρέπει και στον εποπτικό ρόλο και στο ρόλο επισήμανσης και ταυτοποίησης του ρίσκου να έχουμε πάντοτε υπόψη μας και την παγκόσμια πτυχή. Θα έχουμε μία διεθνή προσέγγιση και συνεργασία με διεθνείς ρυθμιστικούς φορείς για να διαμορφώνουμε μία κοινή άποψη όπου είναι αυτό δυνατόν. Αλλά ε, ας πούμε ότι ο ευρωπαϊκός φάρος θα λειτουργούμε σαν φάρος εμείς διεθνώς. Και όπου μπορούμε θα συνεργαστούμε ένεργα ε, με τους σε παγκόσμιο επίπεδο έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, εκμεταλλευτούμε και την εμπειρία μας. Στην Επιτροπή ΑΙΟΣΚΟ σύντομα, ε, πρόσφατα συγγνώμη, όπου είχα μία εμπειρία για την διαχείριση των αγορών OTC ε, διαπίστωσα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο διεθνώς ε, να καταλήξει σε κοινά πρότυπα, αλλά μπορείς να καταλήξει σε κοινού παρονομαστές, στο χαμηλότερο επίπεδο, που πιστεύω ότι αυτός είναι ο στόχος μας ε, στα ρυθμιστικές αρχές. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ο Σβέν. Καλώς ορίσατε και εγώ χαίρομαι, είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος ότι μιλάτε, όχι μόνο η κυρία Ρος μιλά γερμανικά ή μιλάνε οι συνάδελφοι γερμανικά, αλλά ότι η μία συνάδελφος Γαλλίδα μιλά, μίλησε γερμανικά, χρησιμοποίησε μια συναδελφος γαλλιδα μιλησε γερμανικα γλώσσα και μάλιστα ε, δημόσια. Αυτό είναι κάτι το εξαιρετικό από γαλλικής πλευράς. Βεβαίως ιδιωτικά μιλάμε ε, γερμανικά, αλλά για πρώτη φορά δημόσια στο σώμα. Λοιπόν, μέσα στο, στο FSA, στο Financial Services Authority, ήσασταν υπεύθυνοι για τη διεθνής, στο διεθνές τμήμα, στη διεύθυνση διεθνών συναλλαγών και υπάρχει μια, και συντάξατε μια έκθεση η οποία αναφέρεται στη σωστή λειτουργία διεθ, ε, της FSA. Ε, πιστεύω ότι ήσασταν συνυπεύθυνοι για τη σύνταξη αυτού του εγγράφου, αυτή της έκθεσης, όπου χρησιμοποιείται με διαφορετική γλώσσα ε, από αυτήν την οποία επισημούσαμε εμείς στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τις διεθνεί συναλλαγέ, την εποπτεία ε, των χρηματαγορών κλπ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θέση έχετε με αυτή την έκθεση του FSA ε, για ε, την ε, εποπτεία των ε, ευρωπαϊκών και διεθνών αγορών και πού δεν συμφωνείτε, σε ποια σημεία συμφωνείτε με την έκθεση αυτή του FSA και σε ποια διαφωνείτε. Η κυρία Ρος. Όπως σας είπα ήδη και απάντησα προηγουμένως στον προλαλήσαντα, συνεργάστηκα στη σύνταξη αυτής της έκθεσης, δεν το αρνούμε, θα ήταν λάθος αυτό. Όμως είναι ε, ένα έγγραφο το οποίο έχει συγκεράσει ε, μία δέσμη απόψεων μέσα στο FSA. Εάν εγώ προσωπικά είχα συντάξει αυτή την έκθεση, <clears throat> δεν θα είχε αυτό το περιεχόμενο. Θα ήταν διαφορετική. Και για να απαντήσω άμεσα στην ερώτησή σας. Πού συμφωνώ, σε ποια σημεία και πού διαφωνώ ή πού θα είχα επιλέξει μία διαφορετική διατύπωση. Σας λέω το εξής. Εκεί όπου πιστεύω πως το κείμενο όσον αφορά τις Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές ε, ε, αναφέρει σωστά στοιχεία είναι εκεί όπου αναφέρεται στα ευρωπαϊκά, στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και λέει ότι θα, πρέπει, δεν θα, θα υπάρχει ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο, θα υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία για όλες τις ευρωπαϊκές χρηματαγορές. Εκεί δηλαδή όπου υπάρχει η ευρωπαϊκή πτυχή, εκεί συμφωνώ. Εκεί που εγώ θα τα διοτύπανα διαφορετικά, είναι ο ρόλος της ΕΣΜΑ των ο των στελεχών της ΕΣΜΑ σε σχέση με τα στελέχη των εθνικών ε, εποπτικών αρχών. Παρόλο που η ΕΣΜΑ αυτή τη στιγμή είναι ακόμα ένας μικρός ε, φορέας, μια μικρή υπηρεσία, εάν εγώ γίνω εκτελεστική διευθύντρια, θα μεγαλώσει αυτή η υπηρεσία μέσω του κατάλληλη ε, της κατάλληλης τελέχωσης, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στα ευρωπαϊκά συμφέροντα και για να μπορέσει να προσλάβει τους κατάλληλους ανθρώπους. Οπότε πιστεύω ότι τα στελέχη αυτά πλέον της ΕΣΜΑ θα είναι πιο ικανά να δουλέψουν σε ένα πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό ε, πιστεύω ότι όσο το δυνατόν ταχύτερα θα πρέπει να στελεχώσουμε την ΕΣΜΑ με τεχνοκράτες, με τεχνογνώστες ε, και τους, πιο, τα πιο ικανά στελέχη. Και να μην βασιζόμαστε μόνο ε, στη συνεργασία με τους εθνικούς αντίστοιχους φορείς. Ευχαριστώ, η Πρόεδρος. Και τώρα, δεύτερος γύρος ερωτήσεων, ο Μπέρκχαρτ. Ευχαριστώ, κύριε Ρος. Ευχαριστώ ε, που ήρθατε στην Επιτροπή σας. Μου άρεσε πολύ η εισαγωγή σας και δεν θέλω να κάνω ερωτήσεις περαιτέρω για το έγγραφό σας αλλά έχω τρεις ερωτήσεις προς εσάς και θα ήθελα ορισμένες διευκρινήσεις. Καταρχήν, είπατε ότι χρειαζόμαστε στην ΕΣΜΑ ικανούς, ε, ε, ικανά στελέχη για να μπορέσουν να συγκλίνουν οι απόψεις των εθνικών αρχών. Πώς ε, το, μπορείτε να μας το διευκρινίσετε, πώς εσείς βλέπετε τον ρόλο σας. Δηλαδή ε, αντιλαμβάνουμε ότι έχετε επηρεαστεί από την εργασία σας τόσα χρόνια σε Βρετανικό οργανισμό και ε, επίσης είπατε ότι θα διασφαλίσετε και την προστασία του καταναλωτή στα πρέσια της ε, ΕΣΜΑ. Μπορείτε επίσης να μας δώσετε ορισμένα περαιτέρω σχόλια επί του θέματος. Και τρίτον που είναι υποχρεωτικό για αυτή την Επιτροπή και για έναν Ευρωβουλευτή. Σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε πιέσει πολύ για να καταρτιστεί αυτή η αρχή. Πώς βλέπετε ότι θα διαμορφωθεί η συνεργασία σας στο μέλλον με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τα υπόλοιπα και θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ κύριε Βάλς. Η σύγκληση των διαφόρων εθνικών απόψεων θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΣΜΑ και καθορίζεται και γραπτός. Και σαν εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να προβώ στην αναγκαία προετοιμασία κατά τρόπον ώστε οι διάφορες απόψεις οι οποίες εκφράζονται θα πρέπει να συγκεράζονται, να συντονίζονται και έτσι να υποβάλλονται εις την Διοικούσα Επιτροπή για κατά τρόπον ώστε να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τις διαφορές εκ προημίου και να μην υπάρχουν συγκρούσεις διαφορετικών εθνικών απόψεων στη δικούς επιτροπή διότι τότε ε, δεν θα εφαρμόζει την νομοθεσία αυτό το ανώτατο όργανο ε, και θα στρεβλώνεται η δράση του από τις ε, εθνικές διενέξεις. Τώρα, όσον αφορά την Επιτροπή, όπως σας είπα, καταρχήν αυτό το οποίο θα ήθελα είναι να να βελτιώσουμε και να ενοποιήσουμε τους κανόνες πολίσεως ε, και διαχειρίσεως και γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να βελτιώσουμε το νομοθετικό πλαίσιο σαν ρυθμιστές και επίσης θέλουμε να βελτιώσουμε τις γνώσεις του καταναλωτή για το τι αγοράζει ε, να γνωρίζει πού καταλήγει η επένδυση αυτή και τι κίνδυνοι συνεπάγονται στις κινήσεις αυτές και ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν και προϊόντα τα οποία δεν θα έπρεπε να αγοράζει ο απλός πολίτης και πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων του καταναλωτή για επιλογή και ποικιλία και από την άλλη πλευρά προστασία του καταναλωτού που ε, ε, να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι ορισμένα ορισμένα προϊόντα δεν θα καταλήξουν ποτέ προς πώληση στον καταναλωτή. Όσον αφορά αυτά τα οποία είπα προηγουμένως, θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο στη διαδικασία αυτή θα είναι ένας βασικός συνομιλητής μου, διότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε ειλικρινείς και να έχουμε απευθείας συζητήσεις αλλά θεωρώ ότι ε, είστε ένας οργανισμός που θα μπορεί να στηρίξει την ΕΣΜΑ και τον εκτελεστικό διευθυντή της διότι θυμάστε ότι πριν από ένα-δύο μήνες ε, είχατε πιέσει για να υπάρχουν επαρκή σπόροι στη διάθεση αυτής της οργάνωσης οπότε πρέπει να δούμε εάν με τους σπόρους που μας διατίθενται αυτή τη στιγμή θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις απαιτήσει που έχετε από μας. Ευχαριστούμε Πίτερ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε μια υποψήφιο γυναίκα. Είναι δύσκολο στα πλαίσια των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να έχουμε γυναίκες σε τόσο υψηλά επίπεδα. Όσον αφορά τώρα τον ρόλο τον οποίο θα αναλάβετε, την εργασία την οποία θα επιτελέσετε, τι είδου ικανότητε και δεξιότητε μπορείτε εσεί να επιφέρετε. Χρειάζεται μεγαλύτερη ευθύνη, μεγαλύτερη εξουσία, κύρος, μεγαλύτερη ικανότητα όσον αφορά το παγκόσμιο επίπεδο, το ότι θα πρέπει ουσιαστικά να συγκεράσετε όχι μόνο 27 διαφορετικέ εθνικέ εθνιστικές αρχέ, αλλά ότι θα πρέπει ουσιαστικά να έχετε μία παγκόσμια εκπνοβολία. Η CFTC στην Αμερική έχει περίπου 200 ε, εργαζομένους, εσείς έχετε νομίζω περίπου 100 μόνο. Στην Αμερική θα προσλάβουν πολύ περισσότερους, ε, άλλους 400. Ε, Η εργασία την οποία θα επιτελέσετε φαίνεται να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πώς θα καταφέρετε εσείς να επιτελέσετε αυτή την, την περίφημη σύγκληση τι σχέση διοικητική-διαχειριστική θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των ε, εποπτικών αρχών των ε, εθνικών και ποιο ρόλο εσείς θα διαδραματίσετε. Και σε σχέση με τα όσα είπε η Ελίσσα πριν από λίγο, αν δεν κάνω λάθος, στο τέλος της ερώτησής της αναφέρθηκε στην οδηγία για τα hedge funds, AIFM Directive. Suddenly in English, yes. <laughs> Um, I thought that was a bit strange. Um, uh, Ευχαριστώ. Όντως ε, ε, περιγράψατε πολύ καλά τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προσμονές και στις ευθύνες τις οποίες θα μας ε, θα μας ανατεθούν. Θα χρειαστεί μεγάλη εμπειρία και πολλές ικανότητες και πιστεύω ότι αν συγκριθούμε με τη CFTC είναι δύσκολος, δύσκολη σύγκριση διότι ε, αυτή ασχολείται μόνο με τις ε, ε, συναλλαγές για μελλοντική εφαρμογή, τα futures. Επίσης, εμείς θα πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει το σωστό το σωστό προσωπικό και ποσοτικά και ποιοτικά κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις σωστές εμπειρίες στην έσμα των ανθρώπων που είναι απαραίτητοι. Θα πρέπει επίσης η Κοινή Επιτροπή και η Διοικητική Επιτροπή να συνεργάζεται και πιστεύω ότι έτσι θα μπορούμε να υποφεληθούμε συμφωνούμε μεταξύ μας ε, των δυνατοτήτων μας και ε, να εξετάσουμε ε, και τα χρεόγραφα και τις τράπεζες και τη χρηματαγορά και να μην κάνουμε την ίδια δουλειά τρεις φορές και να είμαστε σίγουροι για την ποιότητα των ανθρώπων που θα έχουμε επιλέξει και για τις προτεραιότητες που θα έχουμε καταρτήσει για καθοδήγηση του προσωπικού. Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε τι δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε στο διαθέσιμο χρόνο και γι' αυτό χρειάζεται ε, μία διάφανη ρύθμιση διότι θα πρέπει εσείς σαν νομοθέτες να καταρτήσετε το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσουμε και αν νομίζω ότι δεν θα είναι σωστό τότε αν είμαι επικεφαλής και με επιλέξετε θα έρθω σε εσά για να σας κάνω τα σχόλιά μου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Ε, Είπατε. πριν. Α, αναφέρετε την ΕΣΜΑ ως υπηρεσία. Υπηρεσία. Αρχή. Και μας έχουν πει ότι θα πρέπει να θεωρείτε ως αρχή στα γερμανικά. Αρχή. Εγώ θα έλεγα δεν πρέπει, δεν πρέπει να τη θεωρήσουμε ως παραδοσιακό φορέα από αρχή, αλλά θα πρέπει να είναι μια δυναμική υπηρεσία, μια, ένας δυναμικός οργανισμός, ο οποίος θα, χρησι... θα... θα αντανακλά τις θέσεις τις οποίες υπεραμείνεται. Δηλαδή γιατί ακριβώς προβάλλει, τι ακριβώς κάνει αυτός ο δυναμικός φορέας. Ακριβώς αυτό το οποίο θέλετε κι εσείς να μεταδώσετε με την ομάδα σας, την ομάδα των στελεχών. Ευχαριστώ κύριε Κλίντς, λέει η κυρία Ρος. Ο όρος Behörde έχει λίγο γραφειοκρατική επιβάρυνση ακριβώς. Είναι μια κάπως διοικητική ονομασία, μια γραφειοκρατικής αρχής ή υπηρεσίας. Ας πούμε ότι από απόψεως ε, νομικού προσώπου είναι αρχή η εδμα ε, ή όπως είναι ο τίτλος Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χρηματαγοράς. Αλλά πιστεύω ότι πράγματι θα είναι ένας δυναμικός οργανισμός ο οποίος ε, θα είναι αποτελεσματικός και αποδοτικός ε, και γι' αυτό ακριβώς θα προβάλλει αυτή την ενεργό δυναμική εικόνα. Όσον αφορά τώρα το πρότυπο, πιστεύω ότι θα πρέπει ειλικρινά ε, να το σκεφτώ λιγάκι, αλλά έτσι ε, οι πρώτες σκέψεις, ε, μου επιτρέπετε να σας τις πω, οι πρώτες μου έτσι, ιδέες είναι να δημιουργήσω μία ευρωπαϊκή εποπτεία η οποία θα έχει βάθος όπως λέμε ε, βάθος εννοώ ότι θα, είναι αποτελεσματική και αποδοτική και έναντι εθνικών φορέων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα επιτηρεί την τήρηση και το σεβασμό τη συμμόρφωση με τις οδηγίες. Δεύτερον, ε, θα εξασφαλίζει την διαφάνεια ε, έναντι των βασικών εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων να συμπράξουν και θα προσφέρει μία εποπτεία η οποία θα είναι ανεξάρτητη ε, ε, μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ανεξάρτητη μεν, αλλά μέσα στο ευρωπαϊκό πνεύμα. Ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη ερώτηση είναι από το ΕΛΚΑ, ο Ζαμπόλ Κάρεν. Σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή από την αρχή της παρέμβασής σας. Προέρχομαι από την Ορμανδία και στην Νορμανδία κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που απλώς μιλάνε και σε αυτούς που αναλαμβάνουν και δράση. Πρέπει λοιπόν να μας πείσετε μετά τα όσα είπατε και με τα οποία συμφωνούμε. Γιατί ουσιαστικά και εμείς αυτά θέλουμε να πετύχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θέλουμε πίσω από τα λόγια να κρύβονται πραγματικές δράσεις, πράξεις. Αυτό το οποίο σας ζητάμε αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά να λάβετε δράση και συνήθως δεν γίνεται κάτι τέτοιο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ποιος ξέρει, μπορεί τελικά να επιφέρετε εσείς μια κάποια πολιτιστική επανάσταση. Σας ευχαριστώ. Ε, βεβαίως αντιλαμβάνομαι ουσιαστικά ότι μπορώ να αποδείξω μόνο μέσα των πράξεών μου τι μπορώ να κάνω και εφόσον δεν έχω ακόμη αναλάβει αυτή τη θέση είναι δύσκολο να σας πείσω αλλά <clears throat> μπορώ να σας πω τι έχω κάνει στο παρελθόν και να σας πω πόσο θα ενεργούσα στο μέλλον και εκεί θα ήθελα να αναφερθώ στην άμεση εποπτική εμπειρία εμπειρία την οποία έχω για τα, οι, διάφορ, τους διάφορους χρηματοοικονομικούς ε, ε, οργανισμού, τα χρηματιστήρια και ούτω καθεξής. Σε μια εποχή όπου υπήρχε σύγκληση πολλών εμπορικών συμφερόντων ήταν η εποχή των πρώτων μεγάλων συγχωνεύσεων και υπήρχε μεγάλη πίεση για τις εποπτικές αρχές να υποκύψουν στην εμπορική πίεση και να πούμε ε, εντάξει όλα πάνε καλά προχωρήστε. Εκεί αντελήφθηκα ότι όντως θα πρέπει σαν, επόπτης, ε, σαν εποπτική αρχή να πούμε μέχρι εδώ και μη παρέκει. Δηλαδή θα πρέπει επιπλέον να αποδείξετε ε, ότι αυτά τα οποία υπόσχεστε μπορείτε όντως να τα υλοποιήσετε και αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονίσω διότι αισθάνομαι ότι έκανα κάτι το οποίο ε, εις ε, την θητεία μου της ΕΣΜΑ εάν με επιλέξετε θα μπορέσω και στη συνέχεια να το εφαρμόσω. Ευχαριστούμε Ούτω. Εγώ θα έκανα μία ατμοσφαιρική παρατήρηση και θα έθετα μία ερώτηση. Εσείς ε, είσαστε ε, σαν ε, υποψήφια της City για την θέση αυτή και θα σας έλεγα ότι όποιος έχει τέτοιους φίλους δεν χρειάζεται εχθρούς διότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να ρυθμίσουν φαντάζομαι θα τρομάξουν αλλά σε αυτήν την επιτροπή δεν έχουμε την παράδοση να ακούμε τον τύπο αλλά τις γνώσεις μας και πολύ μου άρεσε αυτό που είπατε μέχρι ότου με επιλέξατε διότι μέχρι στιγμής εσείς έχετε κινηθεί με αγορές για τις οποίες εμείς δεν έχουμε ιδέα για τα παράγωγα εσείς ε, γνωρίζετε ότι ε, επισύουν στους καταναλωτές προϊόντα σαν ε, ζεστά ψωμάκια τα οποία δεν θα έπρεπε να αγοράσει. Τι γίνεται λοιπόν λοιπόν με την ΕΣΜΑ γιατί εμείς πολλές φορές νομίζουμε ότι η οι ε, ε, ρυθμιστέ δεν γνωρίζουν καλά τι χρηματαγορές όπω άλλωστε στην Ιαπωνία με την τωρινή κατάσταση μπορείτε να μας διαφωτίσετε τι είναι τα μέσα τα οποία διαθέτετε και πώ θα τα χρησιμοποιήσετε Σα ευχαριστώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα είναι στις εποπτικές αρχές να έχει τις κατάλληλες πληροφορίες για να μπορεί να κάνει μια, μια ταυτοποίηση και αξιολόγηση του ρίσκου. Αυτές οι προϋποθέσεις πλαίσιο τις οποίες θέσατε πιστεύω ότι θα δώσουν αυτή τη δυνατότητα να συλλέγουμε πληροφορίες μέσω εθνικών εποπτικών αρχών ή και άμεσα απευθείας από χρηματιστηριακές εταιρείες, οικονομικές υπηρεσίες κλπ όχι μόνο για να επισημάνουμε πού προκύπτει ένας κίνδυνος σταθερότητος, αλλά πού υπάρχουν και ποια προϊόντα διατίθενται για εμπορικές συναλλαγές στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτή τη στιγμή ε, για το MRG, για το MIFID συζητούνται διάφορες ε, οδηγίες στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να μην μπορέσουμε επιτέλους να ρίξουμε φως σε αυτό το σκοτάδι σκοτεινό πλαίσιο συναλλαγών. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε περισσότερο πιστεύω το, το διαφωτισμό, τη διαφώτιση την οποία χρειάζεται ο τελικός χρήστης και ο επενδυτής για να χρησιμοποιεί αυτά τα προϊόντα. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε όλο και περισσότερες πληροφορίες. Α, η ισορία, μια χιονοστιβάδα πληροφοριών δεν σημαίνει ότι <clears throat> θα διαφωτίσει και θα ενημερώσει σωστά τον καταναλωτή. Άρα λοιπόν εδώ προσφέρονται θαυμάσιες ευκαιρίες για την ΕΣΜΑ αν και θα είναι πάντοτε εξαιρετικά δύσκολο ως εποπτικό όργανο να είναι συνέχεια κολλημένο πάνω στις αγορές για να παρακολουθεί την καθημερινή δραστηριότητα, τι συμβαίνει, τι τρέχει κλπ. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεργαστούμε με τους ε, stakeholders, δηλαδή με την ομάδα ε, των ενδιαφερομένων, για να μπορούμε μέσω αυτών να λαμβάνουμε επίκαιρες πληροφορίες, ε, αιτήματα και ενδιαφέροντα όλος αυτός ο συνδυασμός των διαφορετικών ε, φορέων πιστεύω μας έχει δείξει ότι πρέπει να προχωρούμε βήμα προς βήμα, προσεκτικά και όχι εντάχει. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε το γύρο των ερωτήσεων και διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά το χρόνο μας, το διαθέσιμο χρόνο. Ε, ε, ευχαριστώ. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον ε, τη συζήτηση και τις απαντήσεις. Αυτό που πιστεύω ότι χρειαζόμαστε είναι ένα ε, ικανό, ε, έμπειρο στέλεχος. Και νομίζω ότι μας δείξατε ότι έχετε αυτές τις ικανότητες, ότι μπορεί να είσαστε αυστηροί, αποτελεσματικοί και δραστήρια αυτό το παιχνίδι της, ε, ε, του, να δακτυλοδεικτούμε ποιος είναι υπεύθυνο για την κατάσταση, ε, ποια υπηρεσία ή αρχή ή φορέας που δημιούργησε ή φταίει για αυτή την κρίση δεν ωφελεί. Νομίζω πάρα πολύ είμαστε όλοι είμαστε λίγο πολύ υπεύθυνοι που δεν είδαμε τι έρχεται κατά πάνω μας, που εθελοτυφλούσαμε. Βλέπω από το βιογραφικό σας ότι μιλάτε κινέζικα, έχετε σπουδάσει μάλιστα την κινέζικη γλώσσα. Ένα συνάδελφός μας μου και πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχετε μια τέτοια γνώση ε, γλωσσική, ε, όπως είναι πολύ χρήσιμο και για τους Βρετανούς να μιλάνε γαλλικά και αντίστροφα. Η κυρία Ρος, ε, μπορώ να σας απαντήσω ε, με μια κινέζικη παραμία που λέει δεν έχει καμία σημασία τι χρώμα έχει η γάτα σας φτάνει να πιάνει τα ποντίκια. Άρα λοιπόν λύσαμε και το γλωσσικό. Η πρόεδρος ε, ήθελα να δώσω στη Βερόνα λίγα λεπτά να ολοκληρώσει γιατί έχουμε λίγο χρονικό περιθώριο. Α, Βίκη. Ε, θα μπορούσατε λίγο να μας διευκρινίσετε κατά την εργασία σας στο FSA τι τεχνικά πρότυπα χρησιμοποιούσατε. Ε, κατά τη διάρκεια του AFM είδαμε ότι υπήρχε μεγάλη διακύμανση και αστάθεια στις χρηματαγορές από άλλα μέρη του κόσμου και γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω τι, ποια ακριβώς πρότυπα θα χρησιμοποιήσετε εσείς και μήπως θα μπορέσετε με τη γνώση σας, της τη γνώση σας κινέζικης γλώσσας να πείσετε και τους Κινέζους να ανεβάσουν το επίπεδο των προτύπων τους στα στις Η κυρία Ρος. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το κάνω αυτό, αλλά ο ορισμός των σωστών προτύπων, των σωστών standards είναι εξαιρετικά ε, σημαντικό διότι θα μας διευκολύνει πρακτικά να δραστηριοποιηθούμε στην διεθνή αρένα, στο, στο, σε διεθνές επίπεδο πρέπει να βρούμε μέσω των κατάλληλων προτύπων ένα κοινό έδαφος για να επισημαίνουμε τους κινδύνους. Ε, σας, ε, στην ΑΙΟΣΚΟ όπου εργάστηκα ε, πρόσφατα ξεκινήσαμε μία μελέτη για τα διεθνή hedge funds. Τι γίνεται λοιπόν σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η πρώτη προσπάθεια που γίνεται καταγραφής σε μία έκθεση των δραστηριοτήτων των hedge funds, διότι πολλές εθνικές αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τι γίνεται με αυτά τα ε, ε, μέσα, με αυτά τα εργαλεία των χρηματαγορών, τα hedge funds και είναι στο σκοτάδι. Εμείς στην Ευρώπη μπορούμε να προωθήσουμε ακριβώς την παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση των hedge funds παγκοσμίως ε, Ιδίω από πλευρά Ασία δηλαδή, βρισκόμαστε ακόμα σε άγνωστο έδαφο. Δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε μεγάλη έλλειψη ε, ενημέρωση. Η Πρόεδρος, ε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που έθεσαν ερωτήσεις. Πιστεύω ότι είναι δίκαιο να δώσουμε στη Βερόνα ένα-δύο λεπτά να ολοκληρώσει την παρουσίασή της. Σε ευχαριστώ Σάρων. Θα ήθελα να σας πω ότι οι ερωτήσεις σας ήταν ιδιαίτερα πλήρεις. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τις ερωτήσεις αυτές. Δεν υπάρχουν σπουδαία πράγματα τα οποία θα μπορούσα να προσθέσω. Επαναλαμβάνω απλώς ότι πιστεύω ότι ε, πρόκειται για μια καταπληκτική ευκαιρία για την Ευρώπη και ελπίζω ότι θα καταφέρετε να μου επιτρέψετε να είμαι και εγώ μέρος της καταπληκτικής αυτής ευκαιρίας και προσβλέπω σε συνεχή συνεργασία μαζί σας και στο μέλλον και αν ε, οποιοδήποτε θέλει να μου θέσει περαιτέρω ερωτήσεις, ακόμα και εκτός της συνεδρίασης αυτής, είμαι στη διάθεσή σας. Προσβλέπω πάντως την ε, έκβαση της ε, συζήτησής σας και των αποφάσεών σας την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ. Right. Thank you very much. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ας α, ε, σταματήσουμε για λίγα λεπτά για να περάσουμε στον επόμενο υποψήφιο.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 Right, παρακαλώ πολύ. Ας περάσουμε τώρα στον δεύτερο γύρο. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε ανάμεσά μας τον Κάρλος Μοντάλβο, επιλεγείς υποψήφιο για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Θα τον ακούσουμε για πέντε λεπτά, στη συνέχεια θα υποβληθούν ερωτήσεις, θα απαντήσει σε ερωτήσεις αυτές πάλι για πέντε λεπτά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να πω άλλα πράγματα, δίνω ευθύ αμέσω το λόγο στον Κάρλος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να έχω τη δυνατότητα να σας μιλήσω για το όραμά μου όσον αφορά την ΕΙΟΠΑ και πώς θα καταφέρω να συμβάλλω στην αρχή αυτή. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω ότι έχουμε μια μοναδική ευκαιρία που μας δίνεται αυτή τη στιγμή να κινηθούμε προς μια ευρωπαϊκή εποπτική αρχή και είναι ευθύνη μας να κάνουμε κάτι τέτοιο. Πώς βλέπω λοιπόν να εξελίσσεται η ΕΙΟΠΑ. Η ΕΙΟΠΑ θα είναι μια νέα ευρωπαϊκή ανεξάρτητη αρχή για τις ασφαλίσεις και τις επαγγελματικέ συντάξεις. Είναι μια νέα αρχή και ξέρουμε ότι οι πρώην επιτροπές level 3 του επίπεδου 3 δεν καταφέραν να επιτελέσουν πλήρως το έργο τους, επομένως έπρεπε να προχωρήσουμε σε μια νέα μορφή αρχής. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για μια πραγματική ευρωπαϊκή εποπτεία. Πρέπει επίσης η ΕΟΠΑ να αποτελέσει το μέσο μέσω του οποίου θα καταφέρουμε να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από οικονομική, τεχνική και πολιτική πλευρά. Πώ θα καταφέρουμε όμω να έχουμε αυτή την οικονομική ανεξαρτησία. Χρειαζόμαστε τον απαραίτητο προπολογισμό και του χρηματοοικονομικού πόρου. Και δεν θα πρέπει βέβαια να δεσμευόμαστε από περιορισμού που θα υποβληθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν θα χρειαστεί και στο μέλλον να έχουμε μια ανεξάρτητη δημοσιονομική γραμμή. Θα πρέπει επίση να είμαστε ανεξάρτητοι από τεχνική πλευρά. Και χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξασφαλίσαμε κάτι τέτοιο. Στι προηγούμενε εκδοχέ του σχεδίου κανονισμού είδαμε ότι υπήρχε μια δυνατότητα να τροποποιηθούν μονομερώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι τεχνικές μονομερείς προδιαγραφές. Πλέον Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Έχουμε μια ξεκάθαρη προσέγγιση με μια ξεκάθαρη συμβολή όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και όλων των συμβαλωμένων μερών. Και αυτό πρέπει να γίνει με εξισορροπημένο, διαφανή τρόπο. Πρέπει από πολιτική πλευρά βέβαια να είμαστε πλήρω ανεξάρτητοι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δίδαγμα από την οικονομική κρίση. Αν δεν υπάρχει πολιτική ανεξαρτησία, οι εποπτικέ αρχέ δεν θα καταφέρουν να επιτελέσουν το έργο του και δεν θα καταφέρει να λειτουργήσει σωστά η ευρωπαϊκή αυτή εποπτική αρχή. Η ανεξαρτησία είναι πάρα πολύ σημαντική σημαντική, αλλά μπορεί να γίνει βάση των δύο βασικών προποθέσεων. Πρώτον, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο λογοδεσία. Και δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο διαφάνεια. Αναφέρθηκα σε μια ευρωπαϊκή ανεξάρτητη αρχή. Πρόκειται λοιπόν για μια αρχή. Δεν είναι απλώς μια λέσχη εποπτικών αρχών. Είναι μια αρχή. Και αυτό γιατί έχει ξεκάθαρες αρμοδιότητες, ξεκάθαρες ευθύνες και θα χρησιμοποιήσει τις αρμοδιότητες της αυτές. Τέλος, ασχολείται με τις ασφαλίσεις και τις επαγγελματικέ συντάξεις. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσει να επιτελεί το έργο της αυτό. Γιατί οι και επαγγελματικέ συντάξεις όχι μόνο από οικονομικής πλευράς αλλά από κοινωνικής πλευράς χρειάζονται ένα συγκεκριμένο έργο, μια συγκεκριμένη αρχή που να ασχολείται με αυτέ. Το ότι ασχολούμαστε βέβαια με τι ασφαλεί και τι επαγγελματικέ συντάξει σε καμία περίπτωση δεν μα εμποδίζει να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία μέσω άλλων κοινών επιτροπών που υφίστανται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προστατεύουμε καταρχά του καταναλωτέ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια εποπτική αρχή. Και όντω αυτό το οποίο έκανα, το πρώτο που έκανα για την ΕΙΟΠΑ ήταν να προσλάβω έναν πολύ σημαντικό εμπειρογνώμονα για τα ζητήματα τη επιτήρηση, τη χρηματοπιστωτική επιτήρηση. Προσπάθησα λοιπόν να έχω έναν συνεργάτη ο οποίος έρχεται πραγματικά από τον κλάδο αυτό που γνωρίζει ακριβώς τι συμβαίνει και τι πρέπει να γίνει. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Χρειαζόμαστε επίσης ένα κοινό εγχειρίδιο κανόνων. Είχα την δυνατότητα να μιλήσω με, τον, με την ομάδα του κυρίου Ντελαροζιέρ και είπα ότι το πιο σημαντικό για μένα, η πιο φιλόδοξη πρόταση που είχε υποβληθεί ήταν ακριβώς αυτό το Single Rule Book, ένα κοινό εγχειρίδιο κανόνων. Συμφώνησε μαζί μου και ενδεχομένως να μην ήταν ε, το πιο δημοφιλές καν επιτρέπεται σεξι μέσο, παρόλα αυτά πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό. Χρειαζόμαστε εναρμόνιση, χρειαζόμαστε συνέπεια και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός κοινού ε, εγχειριδίου κανόνων. Εποπτική αρχή τώρα. Θέλουμε να είμαστε και εμείς ως εποπτική αρχή μέλος του Σώματος Εποπτικών Αρχών, του College of Supervisors. Το ζητήσαμε αυτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, το τόνισε ιδιαίτερα αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην γνωμοδότησή του. Γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να ευθυγραμμίσουμε την ρύθμιση και την εποπτεία με αυτά τα οποία ισχύουν πραγματικά στις αγορές και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να καλύψουμε τόσο την μικροληπτική όσο και την μακροληπτική εποπτεία. Και γι' αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε με την ESRB, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Τέλος, τεχνική συμβουλή στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αρχές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα επιτελέσουμε και το έργο αυτό. Εγώ τι μπορώ να προσφέρω. Έχω ένα ευρωπαϊκό προφίλ. Γεννήθηκα στην Μαδρίτη, ζω στην Φραγκφούρτη, μιλάω τα λεγόμενα ευρωπαϊκά αγγλικά και σίγουρα οι φιλοδοξίε μου και ο προσανατολισμός μου είναι ευρωπαϊκή. Εμπειρία τώρα. Προφανώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά την, το σχέδιο Φεργιότητα 2, Solvency 2, για το οποίο εργάζομαι πάρα πολλά χρόνια, αλλά ασχολήθηκα πάρα πολύ και με το, την ανάλυση της οικονομικής κρίσης και τα διδάγματα τα οποία μπορούμε να, επιτελε, να αποκομίσουμε. Ο Όσκαρ Γουάλτ λέει ότι η εμπειρία ουσιαστικά είναι τα διδάγματα τα οποία αποκομίσουμε από τα λάθη μας. Στο παρελθόν εργαζόμουν στο ΣΕΙΟΠΣ. Γνωρίζω ποιοι είναι οι περιορισμοί του ΣΕΙΟΠΣ. Θεωρώ λοιπόν ότι έχω αποκομίσει και από εκεί τα σωστά διδάγματα προκειμένου να επιτελέσω σωστά το έργο μου στα πλαίσια της ΕΙΟΠΑ. Αυτά μπορώ να προσφέρω εγώ ως υποψήφιος στην ΕΙΟΠΑ, έτσι προσεγγίζω την ΕΙΟΠΑ και τέλος αυτό μπορώ να σας προσφέρω είναι αφοσίωση και σκληρή εργασία. Το μόνο το οποίο ζητώ από εσά είναι η εμπιστοσύνη σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και αρχίζουμε με το γύρο των ερωτήσεων. Ο Ζαν Πολ, καταρχάς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Με ιδιαίτερα προσοχή άκουσα τα, τα όσα είπατε, ιδιαίτερα ικανοποιητικά μου ακούστηκαν και πραγματικά καταδεικνύουν την ευρωπαϊκή σας φιλοδοξία στα πλαίσια της νέας αυτής ευρωπαϊκής αρχής. Αυτό που θα ήθελα να γνωρίζω είναι ότι εφόσον γνωρίζετε το προηγούμενο σύστημα, το ΣΕΙΟΠΣ δηλαδή, θα μπορούσατε να μας πείτε τα νέα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσετε προκειμένου να υλοποιήσετε το σχέδιό σας. Okay? Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Θα απαντήσω στα αγγλικά ή δυνατόν. Ευχαριστώ λοιπόν για την ερώτησή σας. Πράγματι, ήμουν μέλος του ΣΕΙΑ ΟΠΣ και είδα τι ε, περιορισμούς και τι εμπόδια συναντάμε. Το EIOPS είναι τώρα ευρωπαϊκό, ε, μια ευρωπαϊκή αρχή, ευρωπαϊκό νομικό πρόσωπο. Έχουμε διαφορετική δομή, διαφορετική ε, προοπτική πριν από τρεις εβδομάδες μαζί με άλλες εποπτικές αρχές, ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, και άλλους εκπροσώπους ε, πήγαμε στις Ηνωμένε Πολιτείε και συναντηθήκαμε με το NASC, την αντίστοιχη Αμερικανική ρυθμιστική αρχή και διαπιστώσαμε ότι τουλάχιστον στον τομέα των ασφαλίσεων εμείς είμαστε προηγούμεθα, είμαστε πρώτοι, έχουμε καταφέρει πολλά περισσότερα και αυτοί ακολουθούν. Πρέπει λοιπόν και αυτοί ε, να μάθουν από μας ε, και αυτό που καταλάβαμε είναι ότι μία αρχή ε, δεν είναι μόνο ένα νομικό πρόσωπο αλλά είναι και ένα ηθικό ένας ηθικός οργανισμός με ηθικές αρχές αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή η Κομισιόν εργάζεται για ένα, σε μια δέσμη προτάσεων ασφαλίσεων ζωής, ε, με νέες ιδέες. Και αυτό που θέλουμε εμείς είναι να διασφαλίσουμε ότι η, η ΟΠΑ θα ε, μπορέσει να έχει έναν ανεξάρτητο λόγο, να είναι ανεξάρτητος οργανισμός ε, που θα έχει όμως γνώση όλων των προτάσεων που αφορούν τις ασφαλίσεις και τις επαγγελματικές συντάξεις. Ούντο, Κύριε Μοντάλβο, σας καλωσορίζω θερμά. Έχω μία ερώτηση που αφορά την ασφαλιστική αγορά. Είναι μία αγορά με μακροπρόθεσμο ορίζοντα με μακροπρόθεσμους επενδυτές, ο οποίος ε, υποτίθεται ότι ε, πρέπει να καλύπτει βράχει πρόθεσμους κινδύνους και βράχει πρόθεσμα συμβάντα. Και όμως ε, έχουμε την εντύπωση ότι πολλές ε, φορές οι επενδυτές στην ασφαλιστική αγορά επενδύουν με, μακρο, με φιλοδοξίε, πρόθεσμες φιλοδοξίες όπως τα hedge funds και δεν έχουν υπόψη τους τα μακροπρόθεσμα μακροπρόθεσμα ωφέλη και τους μακροπρόθεσμους ορίζοντες. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι μπορεί η, η ΑΙΟΠΑ να ε, προσφέρει έτσι ώστε να προσελκύσει και πάλι τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, αυτοί που θα επενδύσουν για πάρα πολλά χρόνια και δεν θα ενεργούν ως βραχυπρόθεσμοι κερδοσκόποι, όπως τα hedge funds. Ο κύριος Μοντάλβα. Ε, και πάλι. Ε, ευχαριστώ πολύ. Η, η, αγορά ασφαλής, η ασφαλιστική αγορά, συμφωνώ, πρέπει να έχει μακροπρόθεσμους ορίζοντες. Και είμαστε δεσμευμένοι έναντι αυτής της προσέγγισης. Σε προσωπικό επίπεδο βεβαίως και εγώ είμαι ασφαλισμένος για πολλά χρόνια, για το μέλλον. Συμφωνώ λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, διότι τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Ε, τα, τα μαθήματα που, που λάβαμε από την κρίση και σε μια συνάντηση το συζητήσαμε αυτό με τον κύριο Τρισέ, είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της σημερινής κρίσης και της παλαιότερης πριν από 20 χρόνια. Η πρώτη διαφορά είναι ότι δεν έχουμε πλέον τη δυνατότητα βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανταπόκρισης. Πρέπει να αντιδράσουμε ταχύτατα. Το δεύτερο διαφορετικό στοιχείο είναι στην προηγούμενη κρίση υπήρχαν μόνο χαμένοι. Μόνο χαμένοι. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί κερδισμένοι, όμως υπάρχουν και εταιρείε και πολίτες οι οποίοι χάνουν, αλλά υπάρχουν και κερδισμένοι. Τρίτον, δεν πρέπει να ξεχνάμε τι γίνεται ε, σε ε, διεθνείς εταιρείε, όπως στην AIG η οποία εταιρεία διάλεξε να διαλέξει ας πούμε τις εποπτικές αρχές που τη βόλευαν και να αγνοήσει πολλές άλλες ε, και ας μην ξεχνάμε ότι πολλές ε, εποπτικές αρχές δεν είχαν εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Δηλαδή δεν συνεργαζόντουσαν καλά, δεν γινόταν σωστή ανταλλαγή στοιχείων και ενημέρωση. Όταν θέλουμε να επιλύσουμε κρίσεις ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να μπορούμε να βασιστούμε στην σωστή ποιότητα εργασίας των εποπτικών αρχών. Και πρέπει αυτές οι εποπτικές αρχές να είναι πολιτικά ανεξάρτητες Γι' αυτό μόνο μία ισχυρή Ευρωπαϊκή Αρχή μπορεί να έχει την νομιμότητα να δρά ανεξάρτητα και γρήγορα. Εμείς πιστεύω ότι θα, θα, θα, θα, δει, θα φανεί ότι θα προσφέρουμε μια ε, πολύ διαφορετική ε, ε, αντίδραση σε κρίσεις. Κρίσεις θα υπάρχουν πάντοτε, αλλά θα, εμείς θα είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση. Ευχαριστούμε, Σιλβί. Καλημέρα σας ε, κύριε Μοντάλβο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας ξαναβλέπουμε στην Επιτροπή μας. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σε πολιτικό επίπεδο, το οποίο ουσιαστικά ξεπερνά τις δικές σας, το δικό σας προσωπικό προφίλ. Ήμουνα μία από τις ε, εισηγήτριες για το πακέτο μέτρων για την Ευρωπαϊκή Εποπτεία. Αυτό το οποίο θελήσαμε να πετύχουμε είναι να δώσουμε στην Ευρώπη ένα νέο σύστημα εποπτείας, το οποίο θα διαφέρει πάρα πολύ από το σύστημα το οποίο υπήρχε πριν την κρίση. Όταν χρειάστηκε να αποφασίσουμε για τους επικεφαλείς των αρχών αυτών, τοποθετήθηκα λέγοντας ότι δεν θα ήθελα να δούμε τα ε, εκ νέου τα άτομα τα οποία είχαμε στο παρελθόν. Σε καμία περίπτωση δεν καταγγέλω κανέναν, ούτε λέω ότι κάποιος να έκανε καλά τη δουλειά του. Καλούμεθα όμω πάρα πολύ συχνά να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να διέπονται από αυστηρότητα και διαφάνεια. Πώς μπορείτε λοιπόν τώρα εσεί να με πείσετε να επιστρέψω στου Ευρωπαίους πολίτες, στου ε, ψηφοφόρου μου, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί άμεσα από την οικονομική κρίση. Ορισμένοι έχουν χάσει ακόμα και τη δουλειά του. Αυτό είπα και στην κυρία Ρος. Πώς μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια τους, ψηφοφόρου τους ψηφοφόρους μας λέγοντάς τους ότι αλλάζουμε τα πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρώντας τα ίδια άτομα όμως. Και πώς θα καταφέρουμε να τους πείσουμε ότι πραγματικά έχουμε σημειώσει ένα σημαντικό βήμα προς μια πραγματικά πανευρωπαϊκή εποπτεία. Αυτό είπαμε ακριβώς και πριν από λίγο όταν μιλούσαμε με την κυρία Ρος, ότι ε, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να συνεχίσουμε με την ε, ελαφριά αυτή δομή στην νομοθεσία την οποία είχαμε στο παρελθόν όσον αφορά την εποπτεία. Είμαι σίγουρο ότι στη Φραγκφούρτη κάνετε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Πώς μπορώ όμως τώρα εγώ να πείσω τους ψηφοφόρους μου για τη δική σας την επιλογή. Πιστεύω ότι στα πλαίσια μιας οικονομικής κρίσης θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσωπικοί, γιατί αυτό θα επηρεάσει και τον απολογισμό που θα χρειαστεί να κάνουμε στο τέλος. Είμαι ευνοϊκά διακείμενη απέναντί σας, αλλά θα ήθελα και εσείς να με πείσετε για ποιο λόγο πρέπει να σε επιλέξω. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας, λέει ο κύριος Μοντάλβο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η ερώτηση αυτή. Όντως, αυτή τη στιγμή βλέπετε το ίδιο πρόσωπο με αυτό το οποίο γνωρίζετε στο παρελθόν. Αλλά αυτό το οποίο προσπάθησα να κάνω είναι να σας δείξω ότι πραγματικά φιλοδοξώ να αλλάξω τα πράγματα. Θα θυμάστε την πρόταση που υποβλήθηκε για τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχαμε πει ότι θέλουμε μια ανεξάρτητη δημοσιονομική αρχή, έναν εξάρτητο προπολογισμό. Είπαμε επίσης ότι θα πρέπει η επιλογή να βρίσκεται εκτός του συνήθους ευρωπαϊκού καθεστώτος και ότι θέλουμε αυτή τη στιγμή να πετύχουμε τον καλύτερο δυνατό συντονισμό με τις εθνικές εποπτικές αρχές. Είπαμε θέλουμε ότι, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κοινέ τεχνικές προδιαγραφές, καθώς επίσης και ένα κοινό εγχειρίδιο κανόνων. Όλα αυτά όμως θα τίθενται υπό έλεγχο και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, προβλήματα όσον αφορά ζητήματα όπως η εμπιστευτικότητα. Νομίζω ότι ε, έχουμε εντοπίσει τα λάθη του παρελθόντος, θα πρέπει να τονίσουμε περισσότερο πλέον το παρόν και το μέλλον. Θα γίνει την επόμενη εβδομάδα μια σημαντική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πλαίσια της οποίας θα πούμε ότι θέλουμε να είμαστε παρόντες όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι θέλουμε να γίνουμε ως ΕΙΟΠΑ μέλος της παγκόσμιας εποπτικής αρχής για τις ασφάλειες και τις επαγγελματικέ συντάξεις. Επίσης, θεωρώ ότι η εμπειρία που είχα στην Φραγκφούρτη θα πρέπει να σας πείσει για τις ικανότητές μου. Επίσης, θεωρώ ότι ως ΕΙΟΠΑ θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αναλαμβάνουμε κάποιες πρωτοβουλίες Στο παρελθόν είχαμε την ΣΕΙΟΠΣ, αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε εντελώ διαφορετικό λογότυπο για την ΕΙΟΠΑ. Ακόμα και μέσω του διαφορετικού αυτού σήματος, μέσω διαφορετικού λογοτύπου, θέλουμε να δώσουμε το σήμα της αλλαγή. Όντω, στο παρελθόν εργαζόμουν στη ΣΕΙΟΠΣ, τώρα βρίσκομαι στην ΕΙΟΠΑ ή θέλω τουλάχιστον να εργαστώ στην ΕΙΟΠΑ. Αλλά ω εφόσον μιλάμε για μια υποπτική αρχή, ενδεχομένω όντω να έχετε δίκιο όταν λέτε ότι ε, ο άνθρωπο αυτό δεν είναι εξάρτητο, ότι θέλει ουσιαστικά να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τη Ισπανία. Το μόνο που εγώ μπορώ να πω απέναντι στην ε, καταγγελία αυτή είναι ότι θέλω να σας πείσω ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να σας δείξω ότι πραγματικά θέλω να προωθήσω τις αλλαγές και είμαι αφοσιωμένος στο όνομα της αλλαγής. Για να είμαι ειλικρινής, αφήστε το, το λογότυπο. Ας μην αναφέρουμε το λογότυπο. Η πρόεδρος. Η επόμενη ερώτηση από τη Βίκη. Ευχαριστώ. Ως ε, ε, υπεύθυνο της νέας ευρωπαϊκής αυτής αρχής, η ΑΙΟΠΑ, θα στραφούμε σε εσά και για συμβουλές και για το θέμα των ασφαλίσεων, για την προστασία των καταναλωτών και σε άλλα θέματα. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή εξοργίζει τους καταναλωτές στην ασφαλιστική και συνταξιοδοτική αγορά είναι η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εάν μπορεί κάποιος να προσφέρει διαφορετικά ασφάλιστρα αυτοκινήτου σε γυναίκες και διαφορετικά σε άντρες. Βγήκε απόφαση τώρα ότι αυτό δεν γίνεται λόγω ισότητος και γι' αυτό ανέβασε εμένα το κόστος της ασφάλισης του αυτοκινήτου μου πολύ. Ε, ε, Άρα λοιπόν υπάρχουν ακόμα όμως διαφορές στις χρεώσεις των ασφαλιστικών εταιριών. Μπορεί ίσως να πληρώσει ένας άντας παραπάνω στο αυτοκίνητο αλλά λιγότερο στην ασφάλιση ζωής. Λοιπόν ε, ε, ε, υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Έχουμε τώρα ένα χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος ε, του έτους να σκεφτούμε όλα αυτά τα, ε, τις νομικές, ε, νομοθετικές περιπλοκότητες και τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Θέλω λοιπόν να ξέρω πού αδικείται ο καταναλωτής, πού ωφελείται ο καταναλωτής και αν θα έχετε κατά νου τον καταναλωτή στις αποφάσεις Ευχαριστώ για την ερώτησή σας, λέει ο κύριος Μοντάλβο. Ε, εμείς ακολουθούμε μια γενική αρχή την, αρχή της αποφυγής διάκρισης, της μη επιβολής διάκρισης, non-discrimination και για τις ασφαλίσεις και για τις συντάξεις. Αλλά ορισμένες φορές υπάρχουν αποκλήσεις για τεχνικούς λόγους. Όμως, στη ζωή υπάρχουν και άλλα στοιχεία πέραν τεχνικών ε, προσκομάτων που μας οδηγούν σε μία ή στην άλλη απόφαση. Εμείς δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε την ε, απόφαση του δικαστηρίου. Αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι τη σωστή κάλυψη των καταναλωτών. Πώς μπορούμε αυτό να το επιτύχουμε. Σας είπα από τεχνικής απόψεως Υπάρχουν επιχειρήματα που λένε ας κρατήσουμε αυτή την απόκληση, αυτή την εξαίρεση, διότι υπάρχουν αυτοί και αυτοί οι λόγοι. Λοιπόν, για να δούμε αν θα πρέπει να, ε, να διατηρήσουμε ορισμένες εξαιρέσεις ή όχι, πρέπει να εξετάσουμε τις επιπτώσεις. Παραδείγματο χάρη αυτό που έγινε τώρα με την αύξηση του κόστους της ασφάλισης. Δεύτερον, πρέπει να εξετάσουμε ε, τις επιπτώσεις στο γενικό κόστος. Δεν πρέπει να, ένα μέτρο το οποίο αποφασίζουμε να χρησιμοποιείται μόνο για αύξηση του κόστους και του κέρδους ορισμένων ωφελούμενων. Τρίτον, πρέπει να ε, εξετάσουμε ε, εάν συμφωνούν και τα σεσμικά όργανα ε, ή αν υπάρχει περισσότερο περιθώριο διαβουλεύσεων. Αλλά δεν μπορούμε ποτέ να αμφισβητήσουμε βεβαίω μια δικαστική απόφαση. Σας καλωσορίζω κύριε Μοντάλβο. Θα συνεχίσω στα αγγλικά για να μην μπερδευτούμε με τη δική μου γλώσσα τα γερμανικά. Ακόμα και, και τα γερμανικά που μιλούνται στη Φραγκφούρτη πολλές φορές εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω. Ε, και έτσι συνεχίζω στα αγγλικά. Μα, μα αγαπητέ μου Μπούρκαρτ εσύ προέρχεσαι από μια άλλη επαρχία, μια άλλη περιφέρεια. Ελπίζω να μας καταλαβαίνεις. Λοιπόν, συνεχίζω στα αγγλικά. Το Κοινοβούλιο έχει αποφασίσει ότι οι τρεις αυτές ε, αρχές θα πρέπει σαφώς ε, να ωφελούν τον καταναλωτή. Και έχω ένα μακρύ κατάλογο δυσμενών ε, εφαρμογών, δυσμενούς λειτουργίες ασφαλιστικών αγορών. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς θα θεσμοθετήσετε αυτό το, αυτή την προστασία των καταναλωτών τον σε αυτήν την αρχή. Αναφέρεται ήδη ότι θα λανσάρετε καινοτομικά προϊόντα. Αυτό είναι ένα μικρό σημείο, ένα μικρό μέρος των δραστηριοτήτων. Εγώ θα ήθελα να ξέρω τι θεσμικές εγγυήσεις θα προσφέρετε έτσι ώστε η προστασία των καταναλωτών θα παίξει έναν τον σημαντικό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία της αρχής σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην αρχική μου παρέμβαση είπα ότι η βασική μου προτεραιότητα, και ως εποπτική αρχή τουλάχιστον, βασική μας προτεραιότητα είναι η προστασία των καταναλωτών. Όσον αφορά τη δράση την οποία θα αναλάβουμε, πρώτον, έχουμε μια συγκεκριμένη επιτροπή καινοτομία και προστασία των καταναλωτών. Έχουμε τρία άτομα αυτή τη στιγμή στην ΕΙΟΠΑ που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό και αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι άμεσες, ε, άμεσα αποτελέσματα, βραχυπρόθεσμα, αλλά και κάποια αποτελέσματα τα οποία θα έχουν ως ε, στόχο περισσότερο το απότερο μέλλον. Και αύριο στο Παρίσι συνεδριάζει η Επιτροπή αυτή. Θα πρέπει επίση να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ τις ε, καταναλωτικές τάσει οι οποίες παρουσιάζονται και θα πρέπει αυτό να γίνεται από κοινού και με τις υπόλοιπες εποπτικές αρχές. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες καταναλωτικέ τάσεις που διαφορετικά επηρεάζουν διαφορετικούς τομείς τι τράπεζε, τι ασφάλειε κτλ. Είναι σημαντικό να είμαστε σε επαφή με του συναδέλφου μα από του άλλου τομεί. Επίση, θα πρέπει να συλλέξουμε τι βέλτιστε πρακτικέ, οι οποίε ισχύουν αυτή τη στιγμή στι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Αυτό το, η χρηματοπιστωτική παιδεία είναι ένα σημαντικό, εξειδενικευμένο θα έλεγα στόχο, ενδεχομένω να μην καταφέρουμε σε αυτό να πετύχουμε το ανώτερο δυνατό, δυνατό επίπεδο. Όσον αφορά τώρα τι προδιαγραφέ, αυτέ αναφέρονται με απόλυτη σαφήνεια στον κανονισμό. Θέλουμε εμεί πέρα από τι προδιαγραφέ να δημιουργήσουμε και δεσμευτικέ απαιτήσει. Θα πρέπει επίση να καταφέρουμε να προχωρήσουμε στην λήψη των απαραίτητων αποφάσεων. Προκειμένου όμω να καταλήξουμε σε αποφάσει αυτέ χρειαζόμαστε τι κατάλληλε πληροφορίε πρέπει να γνωρίζουμε τουλάχιστον τι τιμή καλούμε εγώ να πληρώσω ως ασφαλισμένος για ποια προϊόντα, για μέσω ποιων υπηρεσιών καλύπτω ως ασφαλισμένος και αν καλύπτονται οι ανάγκες μου πλήρως. Όσον αφορά τώρα την οικονομική κρίση, αυτό το οποίο μάθαμε όλοι είναι ότι δεν πρέπει να αγοράζουμε τα προϊόντα τα οποία δεν καταλαβαίνουμε. Ορισμένοι είπαν ότι δεν θα πρέπει να πολλούν άλλοι τα προϊόντα τα οποία δεν καταλαβαίνουν. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να εξασφαλίσουν ότι κανεί δεν θα πουλάει τα προϊόντα που δεν θα αγόραζε ποτέ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε λοιπόν από τη δική μας την πλευρά μία σημαντική αφοσίωση. Θέλουμε να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό. Έχουμε αναλάβει τη δράση και θέλουμε να προχωρήσουμε στον δρόμο τον οποίο εσείς, ε, στον οποίο εσείς αναφερθήκατε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις δεσμεύσεις αυτές. Εγώ σας μίλησα όμως για την ε, θεσμοθετοποίηση, αν θέλετε, όλων αυτών των πρωτοβουλειών. Τι προπολογισμό θα έχετε, πόσους εργαζομένους θα έχετε στα πλαίσια της αρχής σας. Ο κύριος Μοντάλβο συνεχίζει την απάντησή του. Όπως σας είπα, ξεφύγαμε από την προηγούμενη οργάνωση, η οποία είχε ένα πεδίο ιδιαίτερα περιορισμένο. Έχουμε μια νέα επιτροπή η οποία ασχολείται με τις καταναλωτικές τάσεις και την καταναλωτική καινοτομία, που έχει ως στόχο να προστατεύει όχι μόνο τους καταναλωτές, αλλά και να επιτυγχάνει μια χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τρία άτομα αυτή τη στιγμή ασχολούνται με το συγκεκριμένο αυτό τομέα. Αν σκεφτείτε ότι σήμερα έχουμε 37 συνολικά εργαζομένους, ένας μόλις ξεκίνησε χθε, ήδη ένα 10% ασχολείται με το ζήτημα αυτό ακριβώς, συμμετέχει στην επιτροπή αυτή στην οποία αναφέρθηκα. Ενδεχομένως να μην έχουμε φτάσει το ιδανικό επίπεδο, δεν έχουμε και τους απαραίτητους πόρους ακόμα, αλλά θα υπάρχει και ένας νέος εργαζόμενος ο οποίος θα αρχίσει να ασχολείται ήδη από φέτος με το ζήτημα αυτό. Τώρα, όσον αφορά την, το ποσοστό του προπολογισμού που θα χρησιμοποιήσουμε. Δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Κάναμε κάποιους υπολογισμούς στον προπολογισμό, ο οποίος έχει κατηγοροποιηθεί με βάση συγκεκριμένα κεφάλαια. Για παράδειγμα, πληρωμή προσωπικού, τρέχοντα έξοδα κτλ. Σε κάθε περίπτωση πάντως πιστεύω ότι έχουμε δείξει τη δέσμευση και την αφοσίωσή μας και αυτό φαίνεται ακόμα περισσότερο από το ότι θέλουμε να προωθήσουμε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και όντω μα δεσμεύει για τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε να πετύχουμε στο μέλλον. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την εισαγωγή σας κύριε Μοντάλτο. Έχω τρία ερωτήματα που με ενδιαφέρουν. Καταρχήν, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά το μέγεθος των επιχειρήσεων στην Ευρώπη και αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι εσείς πώς θα κάνετε την αποτελεσματική εποπτεία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ε, έχουν μεγάλες ανησυχίες για την ε, μελλοντική εξέλιξη ιδίως ε, όσον αφορά τις επιπτώσεις Τη ε, της ρυθμίσεως Solvency 2. Επίσης, ε, αν ε, σας επιλέξουμε εδώ στην Επιτροπή, μπορείτε να μου πείτε πόσο θα, πώς θα ξεκινήσετε στη νέα σας θέση, ποιες θα είναι οι κατευθυντήριες γραμμές που θα διαγράψετε στην πρώτη συνάντηση με τους συνεργάτες σας. Και τρίτον, θα θέλαμε ορισμένα στοιχεία ουσιαστικά για τα θερμικά όργανα και εδώ αναφέρομαι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς εσείς δηλαδή διαβλέπετε τη συνεργασία σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Όσον αφορά τα θέματα, ε, κάθε ένα με το ίν, ε, σειρά τους, όσον αφορά τις μικρομεσαίες εταιρείες, η Solvency 2 θα είναι μια σημαντική, η εφαρμογή της οδηγίας Solvency 2 θα είναι πολύ σημαντική, διότι πρέπει να τους αποδείξουμε ότι υπάρχει μια προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο και στο σύστημα ε, υπάρχει ένα παράδειγμα το οποίο ε, ε, συχνά αναφέρω. Αρέσουν τα βιβλία και έχω πολλούς μικρούς βιβλιοπόλους και τους λέγω αν πάρω ένα βιβλίο θέλω μία προστιθέμενη αξία ε, μπορούμε ε, να αντικαταστήσουμε το μικρό αυτό βιβλιοπόλι με το Amazon, όχι βέβαια, το ίδιο είναι και με τις μικρομεσαίες ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν την ίδια σχέση με τους πελάτες τους και άρα οι πελάτες τους θα ενδιαφέρονται, θα παραμείνουν ενδιαφερόμενοι και σχετικά με το Solvency 2 υπάρχει το ίδιο θέμα διότι ε, είδατε ότι αναγνωρίσαμε και ε, λέμε ότι αυτό που ζητάτε είναι πιο, πολύ περίπλοκο θέλουμε να έχουμε ένα πιο απλοποιημένο σύστημα ε, η, η οδηγία αυτή είναι πολύ περίπλοκη και θα πρέπει να μπορέσουμε να τους δώσουμε αυτό που ζητούν από μας όσον αφορά το προσωπικό μας. Ε, το, αυτό που σας είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα άτομα, θα πρέπει να είναι καλοί όσον αφορά την τεχνική βάση τους, θα πρέπει να ενδιαφέρονται για τη δουλειά τους και πρέπει να σας πω με τα μεγάλη υπερηφανία ότι με την ε, ομάδα η οποία έχει καταρτιστεί μπορώ να επιτύχω τους στόχους που έχω θέσει. Τέλος το θέμα των συντάξεων είναι πολύ περίπλοκο και εγώ ξεχνώ συχνά αυτά που ήξερα γιατί είναι τόσο περίπλοκο το θέμα. Άρα θα πρέπει μαζί με τις ακροάσεις τις οποίες θα συμπαρευρεθεί και το Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν έχετε ένα θέμα για τις συντάξεις, ε, για τις χρηματοοικονομικές αναφορές διότι ε, ελπίζουμε ότι θα μπορέσει και το προσωπικό της Ευρώπης και της ε, οργανώσεώς μας να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά, όσον αφορά την παρακολούθηση, εάν θέλουμε να δούμε πώς όσο γίνεται η εμπορία των συνταξιοδοτικών συστημάτων στην Ευρώπη ε, θα μπορούμε να συνεργαστούμε στενά και επικοδομητικά. Ευχαριστώ. Να με ε, συγχωρεί ο Παύλο διότι δεν του έχω δώσει ακόμη το λόγο. Η επόμενη ερώτηση είναι της Ελίζα Φερέρα. Θα μιλήσω αγγλικά για να εξασφαλίσω ότι δεν θα υπάρξει καμία παρανόηση στη μετάφραση. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αναφέρεται στην ανεξαρτησία την οποία η νέα αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει. Και εδώ βλέπουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζουμε την, ε, ε, την, ε, τον κανονισμό είναι ιδιόρυθμος. Θα είστε όντως προασπιστής των ευρωπαϊκών συμφερόντων, είσαστε βέβαιος. Επίσης όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστείτε, υπάρχει μία, ένας τεχνητός διαχωρισμός, αλλά όταν ε, μιλάμε για κινδύνους, οι κινδύνοι προέρχονται από την αλληλοσύνδεση των διαφόρων ε, θεμάτων. Μπορείτε λοιπόν να μας διασφαλίσετε ότι θα συνεργαστείτε με όλους και με το, Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου για να μπορέσετε να προστατεύσετε και τους πολίτες και ε, τους καταναλωτές. Ευχαριστώ. Α ξεκινήσουμε με την ανεξαρτησία. Αναφέρθηκα από την αρχή σε μια ευρωπαϊκή ανεξάρτητη αποπτική αρχή από οικονομική πολιτική ε, πλευρά. Και ότι θα πρέπει να έχουμε ανεξαρτησία όσον αφορά το προπολογισμό μα. Αυτό σημαίνει ότι και οι κυβερνήσει θα πρέπει να μα επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Πώ το εξασφαλίζουμε τώρα αυτό το πράγμα. Πρώτο, με την ποιότητα τη δουλειά μα, Έπειτα με το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχουμε και το οποίο ουσιαστικά αποτελεί έκβαση τη εργασία που κάνατε εσεί εδώ. Τρίτον, το ότι θα έχουμε μία νομική αρχή την οποία εγώ προασπίζω και Τέταρτον, μέσω της δράσης, της ανάληψης δράσης. Αυτό το οποίο είπα και πριν από λίγο είναι ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρούμε ότι η ΕΟΠΑ εκπροσωπεί την ε, γνώμη μιας συγκεκριμένη εθνικής αρχής, για παράδειγμα της Ισπανίας. Θα πρέπει τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα και διαχωρισμένα. Θα πρέπει να έχουμε μια σαφή ανεξαρτησία. Αυτό έχει να κάνει όμως και με τον προπολογισμό που θα έχουμε, με τους πόρους που θα έχουμε και με την ανεξαρτησία που θα μας δώσουν οι εθνικές εποπτικές αρχές. Όντως, στο παρελθόν είμαστε αρκετά εξαρτημένοι. Στα πλαίσια τη ΣΕΙΟΠΣ, για παράδειγμα, υπήρχαν 17 εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών που εκπροσωπώντουσαν στη ΣΕΙΟΠΣ. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει αυτή τη φορά. Ο αριθμό έχει μειωθεί στους 4-5. Όσον αφορά τώρα τις ασφάλειες, τις τραπεζασφάλειε, και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει ο τομέας αυτός, ο ασφαλιστικός τομέας, ο οποίος διαφέρει από τραπεζικό τομέα, να αντιμετωπιστεί εντελώς ξεχωριστά και να υπάρχει και απαραίτητη πυρογνωμοσύνη. Αλλά σαφώς όλοι αυτοί οι τομείς είναι αλληλένδετοι και αυτό φάνηκε και από την οικονομική κρίση. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήρθαμε σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Στιμικού Κινδύνου αυτή την εβδομάδα, όπου προσπαθήσαμε ακριβώς να εντοπίσουμε τους κινδύνους οι οποίοι προέρχονται από τους τρεις αυτού διαφορετικούς τομείς και πώς μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και πώς μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τους πολίτες και τις χώρες. Και θέλαμε επίσης να δούμε πώς λειτουργούν πώς λειτουργεί ο κίνδυνος αυτός ή πώς εκφράζεται σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Επίσης, θέλουμε να αποφύγουμε το ρυθμιστικό αρμπιτράζ, το οποίο το είδαμε να εμφανίζει το σφαινόμενο στο παρελθόν. Θέλουμε να γνωρίσουμε ακριβώς τι συμβαίνει στον κάθε ένα από τους τρεις τομείς. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο, εκτός μικροφώνου. Κύριε Μοντάλβο, εδώ και πολύ καιρό έχετε, ε, ε, εργαστήκατε για το ΣΑΙΟΠ και τώρα αλλάζει βεβαίως ε, φύση, γίνεται EIOPS, Ευρωπαϊκή Αρχή. Μέχρι τώρα ε, έχετε εργαστεί σε πολλές εποπτικές, εθνικές εποπτικές αρχές ε, και τώρα θέλετε εσείς να αναλάβετε την διεύθυνση ως εκτελεστικός διευθυντής ε, πρέπει λοιπόν ίσως να έρθετε σε αντιπαράθεση με εθνικές αρχές να τσακωθείτε μαζί τους ή να συμβιβαστείτε να διαβουλευτείτε με πρώην συνεργάτε, Αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Πώς θα ανταποκριθείτε, πώς θα προσαρμοστείτε σε αυτό το καινούργιο ρόλο. Πιστεύετε ότι θα σας δεχτούν σε αυτό το καινούργιο ρόλο οι παλαιότεροι γνωστοί και συνεργάτες σας, οι οποίοι σα είχαν δύο ισότιμο συνεργάτες, θα σα δεχτούν ω εκτελεστικό διευθύντη τώρα. Ο κύριος Μοντάλβο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι είναι ένας νέος ρόλος και πρέπει να υπάρχει μια νέα αντίληψη. Όπως σας είπα, η... πρέπει να υπάρχει ηθική διάσταση. Ε, στο, παρελθόν υπήρχαν διενέξεις, υπήρχαν διαφορές, ε, υπήρχαν διαφορές μεταξύ ε, του ευρωπαϊκού συμφέροντος και του εθνικού. Αυτά συμβαίνουν πάντοτε, υπάρχουν αντιθέσεις, αλλά ε, το ευρωπαϊκό συμφέρον πάντοτε υπερίσχυε του εθνικού. Εγώ ως νομικός, ως δικηγόρος πρέπει πάντοτε να βρω την σωστή και διαφανή και ξεκάθαρη προσέγγιση. Είτε είναι διαβούλευση, είτε είναι ρύθμιση, επίλυση αντιθέσεων και διαφορών. Πρέπει πάντοτε να είναι ξεκάθαρη στάση μου και ε, πάντοτε να εργαστώ ε, με διαφάνεια. Ε, η προσέγγιση μου πρέπει να είναι διαφανής έναντι όλων των ενδιαφερομένων μερικές φορές ε, ό,τι λέω πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Ε, μερικές φορές σιωπώ, άλλες φορές ε, ξεκαθαρίζω τη θέση μου. δεν γίνεται αλλιώ. Όταν υπάρχει μία αντίθεση, μία αντιπαράθεση, άμα δεν είναι σαφής η θέση σου, δεν μπορείς να τη δικαιολογήσει. Παραδείγματο χάρη, όταν μια μεγάλη χώρα αποφασίσει για μια μικρή, ε, μπορεί να δημιουργηθούν ε, σοβαρές επιπτώσεις. Αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πιστεύω ότι θα με δεχτούν, θα αναγνωρίσουν το νέο μου ρόλο και θα είναι πεπισμένοι ότι μπορώ να εκτελέσω το ρόλο μου σωστά. Η πρόεδρος, ο Πάμπλο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Μοντάλβο που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτά τα οποία καλύπτονται από το, από το Solvency 2 είναι πολύ σωστά, πολύ ικανοποιητικά. Θα ήθελα να ρωτήσω στις αλλαγές που πιστεύετε πρέπει να γίνει στον τομέα των ασφαλίσεων και των συντάξεων ε, σε σχέση με την κρίση. Και επίσης, τι επιπτώσεις ε, θα έχει αυτή η κρίση στις χρηματαγορές, στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Θα σας απαντήσω στα αγγλικά και πάλι, λέει ο κύριος Μοντάλβο δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αποφύγουμε, να γλιτώσουμε τις κρίσεις ή να είμαστε τελείως εξασφαλισμένοι έναντι κρίσεων. Όμως το Solvency 2 ε, βασίζεται σε μια αξιολόγηση οικονομικού ρίσκου και μας προσφέρει ένα εξαιρετικό πλαίσιο άμβλησης κρίσεων και έκτακτων γεγονότων και μας προσφέρει ένα αποτελεσματικό και ε, οικονομικό εργαλείο μέσω ε, διαχείρισης ενδεχόμενων ρίσκων. Αυτό το έχουν αποδεχθεί όλοι οι σεμβαλόμενοι και αυτό το αποδεικνύει και το, η έκθεση QS5. Εάν λοιπόν κάτι συμβεί την Παρασκευή, το Σάββατο λαμβάνω ε, emails, ηλεκτρονικά μηνύματα από το Crisis Task Force, από την Μονάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων, ε, που, εδρεύει, που την δημιούργησε ένας ικανότατος αυστριακός συνάδελφος. Λαμβάνω λοιπόν όλα αυτά τα, τα μηνύματα το Σάββατο και μπορώ να απαντήσω, διότι έχω ήδη τις πληροφορίες, τις έχω αξιολογήσει και μπορώ να κάνω μια πρώτη εκτίμηση. Παραδείγματο χάρη, ε, στην περίπτωση του σεισμού, του τσουνάμι, των πυρκαγιών κτλ. μπορούμε να κάνουμε γρήγορα μια αξιολόγηση. Ε, Επίση, το βαθμό έξεσης όσον αφορά ε, τα, τα χρεόγραφα και την διακύμαση των αξιών και των χρεογράφων στην Ιαπωνική αγορά. Είδαμε ευρωπαϊκές ευρωπαϊκούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ε, ιαπωνική χρηματαγορά και βλέπουμε τι σοβαρές επιπτώσεις είχαν αυτά τα γεγονότα. Ε, από ευρωπαϊκής πλευράς μπορούμε να πούμε ότι οι επιπτώσεις δεν είναι λίαν σοβαρές, είναι υποέλεγχο, ελέγχονται δηλαδή και οι κίνδυνοι είναι τοπικοί, έχουν μια τοπική εμβέλεια, περισσότερο βεβαίως στην Ιαπωνία και εάν χρησιμοποιήσω τώρα το BlackBerry μου, θα έχω άμεση ενημέρωση των χρηματαγορών σήμερα του και των επιπτώσεων. Δυστυχώς όμως πολλές φορές ε, έχουμε δυσάρεστα νέα αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι σλιβερό μεν. Δεν είναι πολλές φορές οι, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία, αλλά πρέπει να μελετήσουμε τις επιπτώσεις στις χρηματαγορέ. Αυτό είναι λυπηρό, αλλά αναγκαίο. Και το κάνουμε αυτό σωστά, συνεχώς και μας, είμαστε δεσμευμένοι στη μείωση του κινδύνου και τη έκθεση σε αυτού. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι κανείς δεν περιμένει να είστε μάντης αλλά κοιτάζοντας τα προηγούμενα λάθη που έχουν γίνει υποθέτω ότι έχετε περισσότερες απαντήσεις από ό,τι εμείς. Ε, ελπίζω ότι το καλό πρόγραμμα που έχουμε δεν θα το, δεν θα το ματιάσουμε και θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε κάνει προσωμιώσεις με εσωτερικά πρότυπα στις επιτροπές και ακόμη δεν είμαι πεπισμένος ότι έχουμε πετύχει. Αλλά εσείς σαν διαχειριστής αυτού του συγκεκριμένου οργανισμού θα πρέπει να τονίσετε την συνεκτική προσέγγιση και να εξασφαλίσουμε ότι όλοι ε, θα πράττουν σωστά ε, το σωστό το καθήκον τους ε, ότι θα υπάρχουν ε, ε, και μετά από τις σοβαρές διαπραγματεύσεις στο Κοινοβούλιο της συνδιαλλαγή και ελπίζω ότι παρόλο που ίσως έχετε αντιταχθεί στις θέσεις μας θα μας βοηθήσετε στο μέλλον και θα έχετε αποτελέσματα αποτελέσματα. Πώς θα επιτύχετε αποτελέσματα βάσει αυτής της συνεκτικής προσέγγισης. Δηλαδή έχουμε μία διεθνή ε, ε, εμπειρία σχετικά με την οδηγία ε, για την επάρκεια των κεφαλαίων 2 Solvency 2. Πώς θα το επιτύχουμε αυτό. Ε, καταρχήν, ας ξεκινήσουμε με την τελευταία σας ερώτηση. Όντως, ο κανονισμός για την επάρκεια των κεφαλαίων, το Solvency II, έχει εξαιρετική φήμη και ε, το, όλοι οι ενδιαφερόμενοι από κοινού καταλήξαμε σε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και επειδή έχω εργαστεί επί του θέματος 10 χρόνια το θεωρώ πολύ καλό όχι όμως ότι δεν επιδέχεται ακόμη με βελτιώσεως είπατε ότι πρέπει να βελτιώσουμε και τα εσωτερικά πρότυπα της προσωμιάσης που κάνουμε και τον τρόπο διεκπαιρεώσεως πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει σωστή εποπτεία αλλά και κίνητρα ε, επίσης ε, το καλό η καλή εσωτερική προσωμείωση θα μπορέσει να μας βοηθήσει βοηθήσει επίσης και να υπάρχει συνεκτικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι δεν είναι όπως σε, άλλες, σε άλλους τομείς ε, όπου υπάρχουν ομάδες που συνεργάζονται με τους ρυθμιστές αλλά επιπλέον ε, έχουμε, ε, έχουμε άτομα τα οποία καθημερινά επιβεβαιώνουν τα εσωτερικά, τις εσωτερικές προσωμιώσεις που καταρτίζουμε. Δηλαδή ήδη τώρα τώρα υπάρχει αυτή η διαδικασία και επιπλέον θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι βελτιώνουμε τον τομέα των εσωτερικών προσωμιώσεων και προσπαθούμε αυτή την παιδεία να την ε, μεταφέρουμε και στην κοινότητα των εποπτών. Να μην έχουμε δηλαδή απλά μέσα, σαν επόπτες πρέπει να δεχθούμε ορισμένα πράγματα που προέρχονται από τους ενδιαφερόμενους και δεν μπορούν να ελεγχθούν εύκολα. Βέβαια έχουμε ήδη αποκομίσει ε, μαθήματα από την τραπεζική κρίση και δεν επιτρέπουμε πλέον μαύρα κουτιά. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα συλλογικά όργανα τα οποία θα επικυρώνουν τα εσωτερικά ε, πρότυπα προσωμιώσεως ε, και ε, γι' αυτό χαίρομαι ότι το προσωπικό της ΕΙΟΠΑ συμμετέχουν στα όργανα αυτά για να μπορούν να συμβάλλουν στην διατύπωση των σωστών αποφάσεων. Και εδώ ίσως ξεπεράσω τα πέντε λεπτά μου πρέπει να σας πω ότι στο πρώτο συλλογικό ασφαλιστικό κολέγιο είχα συμμετάσχει και εγώ σε αυτό το συλλογικό όργανο και εμείς ε, για πρώτη φορά σαν επόπτες ε, μοιραστήκαμε τις εμπειρίες μας για πρώτη φορά. Είναι καλό όμως να γνωρίζεις ποιοι είναι οι συλλομελητές σου και μετά από μερικά χρόνια όταν εργαζόμουν στη χώρα μου συζητήσαμε ε, την διαχείριση του κινδύνου, τους εσωτερικούς ελέγχους, αλλά δεν επαρκούσαν ούτε καν αυτά. Και στη συνέχεια ορισμένα από αυτά τα θέματα τα χρησιμοποιήσαμε και στα κολέγια με τηλέφωνα, με τον εξοπλισμό και πάλι δεν επαρκούσαν και έπρεπε να ξανασκεφτούμε τον όλο τομέα της εκπαίδευσης. Και τώρα έχουμε ένα σύστημα με το οποίο βλέπετε τις ανάγκες της διαχειρίσεως του κινδύνου, των κρίσεων γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει το σωστό πλαίσιο για περίπτωση εκτάκτου ανάγκης και υπάρχουν τεχνητά σενάρια τα οποία θα προσωμιάσουμε για να δούμε τι χρειάζεται για να μπορέσουν να συνεννοηθούν όλοι οι επόπτες και να δουν Ποιο είναι ο ρόλος της και πώς συντονίζει τα διάφορα θέματα. Επίσης δίνουμε αρκετούς πόρους σε αυτά τα όργανα. Υπάρχουν τρεις κατατάξεις, υψηλά, μεσαία και κατώτερα, διότι πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους πρέπει να επιτύχουν. Έχουμε ανεπαρκείς πόρους και πρέπει να γίνει σωστή κατανομή. Πρέπει όμως να υπάρχει σωστή σε όλα αυτά τα εποπτικά κολέγια να έχουμε τη σωστή κατανομή των υπευθύνων και να πιστεύουμε στην ύπαρξη αυτών των οργανισμών διότι σε όλες τις συνεδριάσεις εποπτών υπάρχει στο πρόγραμμα να αναθεωρούμε πώς λειτουργούν αυτά τα εποπτικά όργανα και αρχές Απριλίου θα δείτε ε, το νέο πρόγραμμα δράσης για αυτά τα κολέγια, τα συλλογικά όργανα και θα το δείτε και αυτό διότι θα το έχουμε προωθήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταία ερώτηση, Ίντικα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ επιτρέψτε μου να μιλήσω ουγγρικά. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε να μιλήσω ουγγρικά. Δεν έχω επαρκή χρόνο, διότι είδα ότι είστε πολύ δεσμευμένος και έχετε φιλόδοξα προγράμματα. Αλλά συγχρόνως βλέπω ότι ο χώρος σας είναι πολύ περίπλοκος. Δηλαδή πρόκειται για ένα πολύ συνθετικό χώρο και προηγουμένως το αναφέρατε ότι φτάνουμε στα όρια της αποτελεσματικότητας ε, και ε, ε, φαντάζομαι ότι θέλετε να υπερβείτε τα πλαίσια του παλιού πλαισίου και ε, τώρα υπάρχουν και νέα θέματα τα οποία τίθενται και υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πώς σκοπεύετε να προωθήσετε το θέμα. Αν υπάρχουν τόσες αντιφατικές θέσεις πώς θα τις συντονίσετε διότι και στο μέλλον θα υπάρχουν κίνδυνοι. Πώς θα τους αντιμετωπίσετε. Τι μέσα έχετε για να αναγνωρίσετε τους κινδύνους αυτούς και να τους διαχειριστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Δυστυχώς δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω στα Ουγγρικά θα μάθω όμως και τη γλώσσα αυτή. Όντως, σας είπα ότι οι επιτροπές στο παρελθόν είχαν φτάσει τα όρια τους. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Πριν από δύο περίπου χρόνια, κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου, μια πολύ σημαντική διασυνοριακή οργάνωση συνάντησε πολύ σημαντικά προβλήματα, έπρεπε να ασχοληθώ με αυτό ε, είπα στη γυναίκα μου κάποια στιγμή το Σάββατο ότι αύριο θα μάθεις από τι εφημερίδε ε, ποιε είναι οι αποφάσει οι οποίε ε, ελήφθησαν. Αυτό το οποίο μπόρεσα να κάνω ήταν απλώς να ενημερώσω την αρχή στην οποία βρισκόμουν τότε για το τι μπορούσε να πει, το τι είχε να πει ουσιαστικά το Διοικητικό Συμβούλιο της συγκεκριμένη αυτής ασφαλιστικής οργάνωσης. Νομίζω το παράδειγμα αυτό αποδεικνύει ότι πραγματικά δεν είχα πάρα πολλά μέσα στα χέρια μου. Αυτή τη στιγμή με τη νέα αρχή μπορούμε να καλέσουμε είτε το Διοικητικό Συμβούλιο είτε ίδιο το συλλογικό όργανο, το κολέγιο ή να χρησιμοποιήσουμε την, το μέσο αυτό αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, το οποίο συστήνουμε και θα καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας χωρίς να περιοριζόμαστε στην απλή αποστολή μια επιστολή όπω έγινε στο παρελθόν. Σίγουρα είναι πάρα πολύ αποκαρδιωτικό να πρέπει κανείς να περιγράφει τι μπόρεσε να κάνει κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης όταν δεν είχε σπουδαία μέσα στα χέρια του και όταν το μόνο πράγμα που μπορούσε να κάνει ήταν να στείλει μια επιστολή οι εθνικοί κανόνε και ελάχιστη εναρμόνιση. Μα συμφωνώ μαζί σα. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η πιο φιλόδοξη πρόταση είναι το single rule book, αυτό το κοινό εγχειρίδιο κανόνων. Και εφόσον έχουμε μια κοινή εσωτερική αγορά, θα πρέπει να έχουμε και κοινού κανόνε. Πιστεύω πω ναι. Θα πρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη ευθυγράμμιση και εναρμόνιση. Έχετε για παράδειγμα χώρες στις οποίες έχετε διαφορετικά ασφαλιστικά συστήματα είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να υπάρχει και μια γενικότερη σύγκληση. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πετύχουμε την ελάχιστη αυτή εναρμόνιση μέσω ενός κανονισμού. Γιατί διαφορετικά δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε σε άλλου επιμέρου τομεί υψηλότερη εναρμόνιση. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε του κοινού αυτού κανόνε, θα πρέπει να έχουμε τι ε, νέε ρυθμιστικέ εξουσίε που μα δίνονται μέσω τη νέα αρχή και να καταφέρουμε να συνεργαστούμε και με τι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ επιπτικέ αρχέ όταν και εφόσον αυτέ καταφέρουν επίση να λειτουργούν και ω νομοθέτε και να υποβάλουν νομοθετικέ προτάσει. Πρόεδρος, Νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει τον ε, χρόνο μας. Ένα λεπτό μόνο μπορώ να σας δώσω για να καταλήξετε κάποια συμπεράσματα, για να συνοψίσετε την όλη συζήτηση. Σας ευχαριστώ ναι. πολύ Κοιτάξτε, υπάρχουν τόσα πολλά ζητήματα. Αν επιλέξω ένα από αυτά, νομίζω ότι θα εξαντλήσω το χρόνο που μου δίνετε. Το μόνο που μπορώ να σα δώσω είναι το τηλεφωνικό μου αριθμό και αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο σε απασχολεί, είτε πρόκειται για τι ασφάλειε, είτε πρόκειται για τι συντάξει, μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε και εγώ θα σε όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να σα δώσω μία απάντηση. Είναι πολύ δύσκολο σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να σας εξηγήσω ακριβώς τι πιστεύω και πού θέλω να κινηθώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Ολοκληρώνεται κατά αυτόν τον τρόπο ο δεύτερος γύρος ακροάσεων. Θα κάνουμε πάλι ένα σύντομο διάλειμμα για να περάσουμε στον επόμενο υποψήφιο. Okay, if we could take our seats for round three. Okay, I know, I Η πρόεδρος. Ναι, ξέρω ότι είναι σκληρή η δουλειά σήμερα. Αλλά αν είχατε την καλοσύνη να σταματήσετε τώρα το διάλογο, τις κουβέντες και να εστιάσουμε στην εργασία μας ε, καλωσορίζοντας ε, τον Άνταμ Φάρκας, ο οποίος είναι υποψήφιος για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Ταπεζικής Αρχής. Η διαδικασία, όπως ε, γνωρίζουμε, είναι θα, πρώτα θα έχει ο υποψήφιος πέντε λεπτά στη διάθεσή του να ε, παρουσιαστεί, να μιλήσει. Μετά έχουμε το γύρο των ερωτήσεων και μετά ε, στο τέλος, περίπου ένα λεπτό ξανά, θα έχει ο υποψήφιος το λόγο για να ολοκληρώσει. Ο Άνταμ λοιπόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω την υποψηφιότητά μου ως εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής η ίδρυση, ε, της, ε, Ευρω... του φορέα των Ευρωπαίων ε, Τραπεζικών Εποπτών και η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής ως το ρυθμιστικό όργανο δείχνει ότι η λειτουργία, θα... η λειτουργία αυτής της αρχής θα είναι διασυνοριακή σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια για να εξασφαλίσει την σταθερότητα και τη σωστή λειτουργία των τραπεζών προς όφελο των πολιτών και των, όλων των ενδιαφερομένων. Θα ήθελα ε, να σας παρουσιάσω ορισμένες προτεραιότητες σε τέσσερις τομείς όπου χρειάζεται να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος ε, και να δοθούν ε, αρμοδιότητες πρόσθετες στην EBA, σε αυτή την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή για, θέλοντας να δημιουργήσουμε νέους κανόνες για την τραπεζική αρχή στην Ευρώπη θα πρέπει καταρχάς να εφαρμόσουμε το CRD4 να υλοποιηθεί λοιπόν ε, ε, αυτό το, το πλαίσιο για τη διαχείριση κινδύνων. Όσον αφορά τώρα την εποπτεία και την λειτουργία των ε, ρυθμιστικών αρχών, έχω τρεις προτεραιότητες. Πρώτον, η αξιόπιστη εκτέλεξη, εκτέλεση stress test, δηλαδή δοκιμών αντοχής των τραπεζών. Δεύτερον, βελτιώσεις στο κολεγιακό σώμα εποπτών, στο διατραπεζικό σύστημα και τρίτον να ανυψώσουμε το ρόλο της EBA σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, για την προστασία των καταναλωτών. Στον τρίτον αυτό τομέα, τον οποίο εγώ καθορίζω ως προτεραιότητα αποφυγής συστημικών κινδύνων στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό πλαίσιο, είναι ένας ρόλος κλειδί εδώ σε αυτό τον τομέα που θα παίξει η EBA. Δηλαδή θα παίξουμε έναν δραστήριο ρόλο στη προσπάθεια να αποφύγουμε συστημικές κρίσεις ε, διασυνοριακά. Και δεύτερον, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ε, να ενισχύσουμε τις εργασίες των κοινών επιτροπών μεικτών επιτροπών για να ε, προσφέρουμε μια καλύτερη διατομεακή εποπτική ε, εργασία. Ε, και Τώρα, στο εκτελεστικό, εκτελεστική προτεραιότητα θα πρέπει να αρχίσουμε πολύ ήπια ε, με την εφαρμογή των νέων κανόνων λειτουργίας, δεδομένου ότι είναι μια καινούργια αρχή και πρέπει να, να υλοποιηθούν ο, ο, ο κανονισμός λειτουργίας ταχύτατα για να μπορέσουμε να εργαστούμε επιτυχώς. Έχουμε ένα σημαντικό έργο συλλογής ε, και διαχείρισης δεδομένων δεδομένα τα οποία θα είναι επαρκή και αξιόπιστα και θα προέρχονται από τον τραπεζικό ευρωπαϊκό κλάδο και τα οποία δεδομένα θα μπορούμε να αναλύουμε και να μελετάμε για να, προσ... για να συντάσσουμε προτάσεις και συστάσεις στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν μια ισχυρή δύναμη υποστήριξης ε, για την δημιουργία της CBA και έχει υποβάλει προτάσεις ε, για ε, την λειτουργία και την μελλοντική εξέλιξη του, της αρχής. Σας διαβεβαιώνω ότι θα, κάνω κάθε, θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια να δώσω την ευκαιρία στην EBA να χρησιμοποιήσει ως ανεξάρτητη αρχή τις νέες αρμοδιότητες, την καινούργια της ισχύ για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών και εκείνων που διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή πολιτική. Θα Έχω πρόθεση να επικοινωνούμε τακτικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ε, να μπορέσω να απαντήσω στο πώς έχουμε μεταφέρει τις προσδοκίες, πώς έχουμε υλοποιήσει τις προσδοκίες του σώματος ε, σε προγράμματα. Ε, προσβλέπουμε μεγάλη χαρά στη συνεργασία μου με τα στελέχη της EBA για να, για να προωθήσω το έργο της CBA και στηρίζουμε και στην, στην Επιτροπή σας. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Πρώτος γύρος των ερωτήσεων από τον Ζαν Πολ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Φάρκας. Δεν θα είμαι πολύ πρωτότυπος και ε, θα σας ζητήσω να με, ε, να, ε, να με συγχωρήσουν όσοι παρακολουθούν από το πρωί τις συνεντεύξεις αλλά θα ήθελα να ξέρω και από εσά από τη σκοπιά του Κοινοβουλίου πώς προβλέπετε ότι ε, θα επιβληθείτε και ε, θα μπορέσει να αυξηθεί το κύρος της, ε, της αρχής της οποίας θα είστε επικεφαλής. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ελπίζω ότι είναι ανοιχτό το μικρόφωνο μου. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο θα εξασφαλίσουμε ότι η αρχή ε, θα είναι σωστά εγκαθιδρυμένη και ε, θα γίνει σεβαστή θα βασίζεται στις νέες εξουσίες με τις οποίες θα λειτουργήσει ε, αυτή η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή διότι χωρίς να αναφερθώ στις λεπτομέρειες θέλω να τονίσω τρεις τομείς. Καταρχήν η Τραπεζική Αρχή θα μπορέσει να καταρτήσει ρυθμιστικές προδιαγραφές. Με συγχωρείτε, ίσως δεν ήμουνα σαφής. Εγώ μίλησα για την δικιά σας, για, την δικιά σας, για το δικό σας κύρος, για τη δικιά σας προσωπική επιρροή για να εγκαθιδρύσετε και να στηρίξετε αυτή την αρχή. Με συγχωρείτε αν στραβοκατάλαβα. Σαν εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής ε, θα διασφαλίσω ότι η αρχή αυτή θα λειτουργήσει ε, βάσει σε πολύ υψηλό επαγγελματικό επίπεδο και ότι δεν θα επηρεάζεται από τις κυβερνήσεις, από τις εθνικές αρχές, από τα θεσμικά όργανα, αλλά θα εφαρμόσει την εντολή να εξασφαλίσει χρηματοοικονομική σταθερότητα και θα χρησιμοποιεί την κρίση της και τον κοινών ε, για να διατυπώσει ε, ε, συμβουλέ για την πολιτική ή να διαμορφώσει προδιαγραφές. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Κύριε Φάρκας, με μεγάλη χαρά σας ακούμε σήμερα. Εμείς ζητήσαμε ηγεσία, ηγεσία σε αυτή τη θέση και θέλουμε κάποιον ο οποίος πραγματικά θα είναι ο άριστος διότι μέρος της ευθύνης του είναι να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της μηχανής με την κατάλληλη ταχύτητα. Υπάρχουν τέσσερα ζητήματα που ανακύπτουν εδώ. Μας είπατε τους στόχους σας, τις προτεραιότητες, το όραμά σας και την εκτέλεση την ε, υλοποίηση των προθέσεων. Η παρουσίασή σας αναφέρθηκε στο πώς θα ανταποκριθούμε στα τεστ αντοχής των τραπεζών, πώς θα ανταπεξέλθουμε σε αυτή την κρίση την τραπεζική. Όμως η τραπεζική αρχή αυτή πρέπει να συντονίσει και τις κατάλληλες ε, λύσεις. Δηλαδή θα πρέπει φέτος να προετοιμάσετε την πρώτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι θέλετε να αναφέρει αυτή η έκθεση, πώς θα διαμορφώσετε αυτή την πρώτη έκθεση. Επίσης θα θέλαμε να ξέρουμε το πολιετές πρόγραμμα της CBA με τις προτεραιότητες της αρχής. Επίσης υπάρχουν διάφορες ε, αρμοδιότητες που αναφέρεται, καταρχάς οι ευθύνες ε, προς τον ιδιωτικό τομέα. Π.χ. θα ήθελα να ξέρω ε, τι ακριβώς σημαίνει αυτή η ανάληψη ευθυνών για σας. Πώς τις, πώς ερμηνεύετε. Ο κύριος Φάρκας. Πιστεύω ότι υπάρχουν ε, ε, μου θέσατε τρία σαφή ερωτήματα. Πρώτον, τι θα περιέχει αυτή η πρώτη έκθεση. Πώς θα διαμορφωθεί. Νομίζω ότι στον κανονισμό της CBA λέει σαφώς ποια είναι η εντολή και ποια είναι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της CBA έναντι των ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών συστημάτων. Ο κανονισμός εργασίας και η έκθεση θα πρέπει να οικοδομηθούν επί τη βάση αυτών των ε, διατάξεων, του κανονισμού λειτουργίας, ε, του κανονισμού σύστασης. Και επίσης βάσει αυτής της εντολής θα αξιολογηθεί και η απόδοση της EBA. Ως εκτελεστικός διευθυντής λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω να επισημάνω τις προτεραιότητες που προκύπτουν από τον κανονισμό και θα μετρήσω τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματα της CBA σύμφωνα με αυτές τις ε, εντολές του κανονισμού στο πρόγραμμα εργασίας το οποίο ναι, θα προταθεί από το σώμα της τραπεζικής αρχής και θα εγκριθεί από, το, από την αρμόδια η εποπτική αρχή θα καλύπτει τις βασικές προτεραιότητες των δύο-τριών επόμενων χρόνων. Αν έχουμε κατά νου την υλοποίηση του CRD4, ε, θα ε, κατανοήσουμε ότι είναι ένα πολιετές μεγάλο, βαρύτατο πρόγραμμα. Ε, δεν είναι μόνο ετές, δεν είναι ετήσιο. επίσης για ε, την ε, αξιολόγηση συστημικών κινδύνων. Είναι ένα έργο με μακροπρόθεσμη πρόπτικη, όχι μόνο ετή. οι προτεραιότητες λοιπόν θα είναι κρίσιμες προτεραιότητες για το πολιετές πρόγραμμα εργασίας. Τώρα, ε, ποιες είναι οι δικές μου ευθύνε συγκεκριμένα ως εκτελεστικού διευθυντή στο να ε, υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα, αυτό πάλι καθορίζεται σαφώς το κανονισμό. Είναι μία λειτουργική ευθύνη. Ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να εξασφαλίσει την επαρκή και ε, βέλτιστη στελέχωση του φορέα ότι την υλοποίηση της σωστής ροής εργασιών και την ε, ε, τα, αποτελέσματα, την υλοποίηση των, των προγραμμάτων, την παραγωγή δηλαδή αποτελεσμάτων. Ε, θα στηριχθούμε σε επαγγελματικό προσωπικό το οποίο θα έχει όλες τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις θα συντονιστούμε με τους stakeholders του τομέα, τους ενδιαφερόμενους δηλαδή και θα γίνει πλήρης αξιολόγηση των εσωτερικών μας λειτουργιών. Ως προς την ανεξαρτησία της αρχής θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Ανεξαρτησία της εντολής. Στο άρθρο 52 αναφέρεται αυτό. Απάντηση. Η ανεξαρτησία όσον αφορά τουλάχιστον τον εκτελεστικό διευθυντή τι σημαίνει στην καθημερινή μου δραστηριότητα δεν θα μπορούν να γίνουν δεκτές οδηγίες συστάσεις από άλλα συμβαλόμενα μέρη, κυβερνήσεις, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δεν θα πρέπει να ασκείται πίεση από τον ιδιωτικό τομέα ή από τον βιομηχανικό κλάδο. Ανεξαρτησία όμως επίσης ε, συνεπάγεται και τον ε, επαρκή αριθμό πόρων, επαρκή ποσότητα πόρων για την αρχή αυτή, προκειμένου να είναι σε θέση να επιτελεί με ανεξάρτητο τρόπο τα καθήκοντά της. Και σαφώς βέβαια ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να προασπίζει την ανεξαρτησία και βέβαια να προσπαθεί με κάθε τρόπο να εξασφαλίσει το απαραίτητο επίπεδο πόρων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Η Σιλβή για την επόμενη ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Φάρκας. Όπως το είπε και ο Ζων Πολ Γοζές, είμαστε υποχρεωμένοι να επαναλαμβάνουμε αυτά που έχουμε ήδη πει, αλλά με εσάς έχουμε ένα νέο πρόσωπο και ένα άτομο που έρχεται από μία χώρα που έχει είχε δυσκολίες δημοσιονομικές και ε, ε, δεν ε, εξετάζεται όμως αυτή τη στιγμή, δεν είναι στο προσκήνιο των προβλημάτων. Ήθελα λοιπόν να σας πω σχετικά με την απόφαση που ελήφθη από τους 17 την περασμένη εβδομάδα βάσει της, του του ανταγωνιστικότητος όπου συνεφωνήθη κατόπιν προδρομής της Γαλλίας και της Γερμανίας το Φεβρουάριο. Χρειαζόμαστε λοιπόν εθνικά, εθνικές αποφάσεις ε, για να βγούμε από την ε, κρίση και θα ήθελα να ξέρω πώς εσείς αντιμετωπίζετε αυτή την κατεύθυνση που δίνουν ε, οι κυβερνήσεις των κρατών για αυτούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον τραπεζικό χώρο ε, από το πρίσμα των ε, αρμοδιοτήτων σας σαν εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχές για να μπορέσει να εφαρμοστεί εφαρμοστεί η αρχή της εσωτερικής αγοράς να μην υπάρχουν μόνο τοπικές τράπεζες διότι υπάρχουν πολλές τράπεζες οι οποίες εδρεύουν σε μία χώρα και δραστηριοποιούνται σε μία άλλη. Νομίζω ότι όντως ε, είναι πολύ λεπτό και πολύ δύσκολο θέμα αυτό διότι ε, όντως θα έπρεπε να εξετάζουμε την αρχή αυτή από την προοπτική των τραπεζών και αυτός, ε, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Όσον αφορά την άσκηση των ε, stress test και των θεμάτων που εξετάστηκαν είναι το θέμα του ο κινδύνου των κρατών από πλευράς τραπεζικής. Αυτό το οποίο θα ήθελα και θα προσπαθούσα θα ήταν οι δοκιμές αυτές, τα stress test των τραπεζών να είναι αξιόπιστες και για τις τράπεζες να ξέρουν ότι μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα και μεταξύ τους και στα, στα μάτια ε, των επενδυτών, των των πολιτών και τα λοιπά. και επίσης αυτά τα stress test θα πρέπει να είναι αξιόπιστα για τους επικεφαλής των κρατών και ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα προσπαθούσα λοιπόν να δω πώς μπορούμε να επιτύχουμε αξιοπιστία, πώς αυτά τα stress test μπορούν όντως να εκπληρώσουν το στόχο για τον οποίο έχουν επινοηθεί. Και εδώ το βασικό θέμα είναι πώς θα εξετάσουμε για αρνητικές δυσκολίες, προβλήματα ή σενάρια κινδύνου σε ορισμένα κράτη και σε ορισμένα χρεόγραφα που έχουν οι τράπεζες στα βιβλία τους στο πνεύμα το οποίο διέπει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πώς θα δοκιμάσουμε και θα κάνουμε το stress test των στοιχείων των βιβλίων των τραπεζών, του, της περιουσίας των τραπεζών που θα πρέπει να αντισταθούν σε δονήσεις σε, σε περίπτωση που υπάρξουν καταστροφικά σενάρια που υλοποιούνται. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να να ε, επιλέξω μία πιο αυστηρή ε, προσέγγιση, μία πιο ε, ανοιχτή υποβολή και αποκάλυψη των στοιχείων όλων και να δω τις θέσεις των τραπεζών αυτών κατά τρόπον ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε κάθε περίπτωση. Εάν δηλαδή το θέμα αυτό χρειάζεται να επανέλθει στο επίπεδο του Συμβουλίου, δηλαδή των αρχηγών κρατών, πιστεύω ότι με τη διαβούλευση ή μετά από διαβούλευση με το Προεδρείο και με την το Εποπτικό Συμβούλιο θα μπορέσει η αρχή μου να επαναφέρει προς συζήτηση το θέμα και εάν θεωρώ ότι είναι αναγκαίο δεν θα διστάσω να το ζητήσω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω ένα λεπτό ερώτημα αυτή τη στιγμή γιατί ε, ο εκτελεστικός διευθυντής είναι μια θέση ιδιαίτερα υψηλή και δεν πρόκειται για μια θέση μόνο επαγγελματική αλλά και πολιτική. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και αλλού όταν προσπαθούμε να δούμε πώς ε, οι νέες αυτές εποπτικές αρχές, όχι μόνο η EBA δηλαδή, αλλά η και η ΟΠΑ θα πρέπει να συσταθούν όταν συζητούσαμε τον όλο σχεδιασμό τους, Είπαμε ότι από τη μια θέλουμε να έχουμε συντονισμένους κανόνες κοινούς, αλλά από την άλλη θέλουμε να υπάρχει και ένα κάποιο περιθώριο για μια ανεξάρτητη ανάληψη πρωτοβουλειών από τις εθνικές εποπτικές αρχές. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η EBA θα είναι σε θέση να επιβάλλει δεσμευτικούς κανόνες στις εθνικές εποπτικές αρχές, αλλά παράλληλα οι εθνικές εποπτικές αρχές θα είναι σε θέση να επιβάλλουν το δικό τους όραμα όσον αφορά τη λειτουργία της ε, EBA. Και αυτό φαίνεται άλλωστε από τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επομένω, ε, ποιο είναι ο αρχηγό σε συγκεκριμένη περίπτωση, εσεί είστε αρχηγό των Εθνικών Εποπτικών Αρχών ή είστε υπό την καθοδήγηση των Εθνικών Εποπτικών Αρχών. Ξέρω ότι η ισορροπία είναι πολύ λεπτή και ότι ε, θα πρέπει να έχετε πολύ καλές πολιτικές δεξιότητες πέρα από τις πολύ καλές επαγγελματικές δεξιότητες που σαφώς έχετε για να πετύχετε τη λεπτή αυτή ισορροπία απάντηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όντως, οι σχέση στην οποία αναφερθήκατε είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη ανάμεσα δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ή σε μια, ανάμεσα σε μια οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή και τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές. Νομίζω ότι έχετε δίκιο όταν λέτε ότι όσον αφορά την ε, διακυβερνητική διάσταση της EBA, έχουμε τους επικεφαλείς των Εθνικών Εποπτικών Αρχών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό αληθεύει. Αλλά σύμφωνα με τον κανονισμό, οι εθνικές αυτές εποπτικές αρχές δεν θα εκπροσωπούν πλέον τα κράτη-μέλη, τα συμφέροντα των κρατών μελών από τις οποίες προέρχονται, αλλά θα πρέπει να υιοθετούν αποφάσεις προς το συμφέρον του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι έχουμε τώρα μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τα όσα συνέβαιναν στο παρελθόν στις επιτροπές του επίπεδου 3 όπου ε, στο παρελθόν είχαμε επιτροπές που εκπροσωπούσαν ουσιαστικά εποπτικές αρχές από συγκεκριμένε χώρες που ουσιαστικά εκπροσωπούσαν τι χώρε αυτέ, ενώ εδώ έχουμε του επικεφαλεί μεν των επιπτωτικών αρχών που λειτουργούν και συζητούν προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην καθημερινή μα τώρα εργασία, ο καονισμό λέει ότι ε, σαφώ οι εθνικέ εποπτικέ αρχέ εξακολουθούν και έχουν πρωταρχικό ρόλο. Αυτό λέγεται ξεκάθαρα. Ωστόσο όμως βλέπουμε ότι η EBA θα έχει την ε, δυνατότητα να έχει συγκεκριμένα μέσα, σημαντικά μέσα, προκειμένου να επιτύχει συνεκτικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναλάβει ακόμα και δράσει σε έκτακτε καταστάσει, πράγμα το οποίο δεν προβλεπόταν στο παρελθόν, δηλαδή στι level 3 committees. Να, αναφέρω επίση ότι η EBA θα αναλάβει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την εφαρμογή και την επινόηση κανόνων, τεχνικών προδιαγραφών. Η EBA επίσης θα έχει σημαντικές αρμοδιότητες όσον αφορά την περίπτωση εκείνη που θα εντοπιστεί κάποια παραβίαση κοινοτικών κανόνων από κράτος μέλος, η EBA επίσης θα έχει σημαντικές αρμοδιότητες όσον αφορά την παρακολούθηση της λειτουργίας των colleges, των συλλογικών αυτών οργάνων εποπτικών αρχών και επίσης η EBA θα έχει σημαντικές αρμοδιότητες όσον αφορά την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επίσης θα έχει και κάποιες αρμοδιότητες διευθέτησης διαφορών. Σαφώς ε, η διαδικασία θα είναι πολιτικής φύσης, αλλά μετά την ε, πρώτη αντιμετώπιση ε, διενέξεων, την πρώτη διευθέτηση διαφορών, πιστεύω ότι θα ξεκαθαριστεί το τοπίο στα πλαίσια των συμβαλωμένων μερών που συμμετέχουν. Επίσης, οι οργανώσεις οι οποίες συμμετέχουν στην EBA θα πρέπει να υποβάλουν συγκεκριμένε επαγγελματικές γνωμοδοτήσεις και αν υπάρχει μία κάποια απόφαση η οποία θα αντίκειται στην ε, δικλίδα ασφαλείας η οποία προβλέπεται στον κανονισμό της EBA, πάλι εναπόκειται στην EBA να πάρει την τελική απόφαση, να κρίνει αυτή δηλαδή ποια απόφαση θα πρέπει να ακολουθηθεί. Κάτι ακόμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει είναι η προστασία των καταναλωτών. Έχουμε νέες αρμοδιότητες ως προς αυτό και σύμφωνα με την ανάλυση που κάνει των αγορών, αν εντοπιστούν μη θεμητές πρακτικές από επιχειρήσεις σε ορισμένα κράτη-μέλη μπορεί η EBA να αναλάβει δράση και ακόμα να φτάσει μέχρι το σημείο να περιορίσει τις εμπορικές δραστηριότητες ή την πόλη συγκεκριμένων προϊόντων υπηρεσιών από συγκεκριμένε επιχειρήσει. Νομίζω ότι αυτό πραγματικά τροποποιεί πάρα πολύ σημαντικά τη σχέση η οποία υπάρχει μεταξύ τη CBA και των εθνικών εποπτικών αρχών. Πρέπει να σα πω ότι όσον αφορά την επαγγελματική εμπειρογνωμοσύνη, όσον αφορά την συλλογή των καλύτερων δυνατών πρακτικών, η EBA θα είναι στην καλύτερη δυνατή θέση προκειμένου να συντονίσει και να χρησιμοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη η οποία έχει συσσωρευτεί στις εθνικές εποπτικές αρχές. Ευχαριστώ. Ο Σβέν. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Θα μιλήσω αγγλικά. Δεν χρειάζονται τα ακουστικά σας, κύριε Φάρκας. Λοιπόν, η ομάδα μας ανησυχεί ιδιαίτερα βλέποντας τις πολύ ισχυρέ πιέσεις ε, από τον τραπεζικό τομέα πάνω στους νομοθέτες και τις ρυθμιστικές αρχές να τους λένε συνέχεια ε, οι τράπεζες μην το παρακάνετε, μην το παρακάνετε λόγω των επιπτώσεων της ε, χρηματοοικονομικής κρίσης ταυτόχρονα τα μπόνους και τα μερίσματα και η διανομή αυτών Ε, λέμε ότι θα υπαχθούν στις ε, νέες ε, τραπεζικές ρυθμίσεις. Θέλουμε την επιβολή αυστηρών κανόνων για τα μπόνουσες και για τις αμοιβέ. Η αρχή σας θα έχει το ρόλο να ελέγχει εάν οι εθνικές εποπτικές αρχές υλοποιούν και εφαρμόζουν αυτούς τους νέους κανονισμούς τι θα κάνετε εσείς για να ελέγξετε ε, αυτό το, το θεσμό των πόνους ώστε να είναι δίκαιος και σε μητός. Ο κύριος Φάρκας, πιστεύω ότι η EBA θα έχει την ισχύ ε, και βεβαίως ε, το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει και την ευθύνη να παρακολουθεί την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων είτε είναι κεφαλογικές απαιτήσεις είτε είναι κανόνες και συστάσεις για τις αμοιβέ και τα μπόνους. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έχουμε την υποχρέωση ε, για μία αναθεώρηση, να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα πάνελ με την ε, ευθύνη της παρακολούθησης και ε, ε, ανασκόπησης της κατάστασης σε τακτικά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα της κατάστασης και να μπορούμε να συγκρίνουμε τις, τα διάφορα στοιχεία εν συνεχεία να συζητήσουμε τα πορίσματα το Διοικητικό Συμβούλιο και αν χρειάζεται να, λάβουμε, να αναλάβουμε δράση ε, εάν διαπιστώσουμε ότι αυτοί οι κανονισμοί υποχρεωτικοί δεν τηρούνται. Η πρόεδρος, ε, ο Σβέν ξανά. Ναι, ακριβώς για τις αμοιβέ και τα μπόνους Σημερίζεστε την ε, ανησυχία την οποία εγώ εξέφρασα ότι δεν υλοποιούνται, δεν γίνονται σεβαστοί οι κανόνες και τι θα κάνετε γι' αυτό. Ο κύριος Φάρκας, ναι, ναι, ναι, συμμερίζουμε τις ανησυχίες σας ότι υπάρχει έντονη πίεση κατά της ε, επιβολής αυτών των νέων κανόνων και επίσης υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην ερμηνεία αυτών των κανόνων στα χέρια των εθνικών εποπτικών αρχών. Αυτό που μπορώ να πω ότι είμαι έτοιμος να αναλάβω δράση εάν χρειάζεται εφόσον έχει γίνει μία μελέτη και ανάλυση το, της κατάστασης και καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται δράση θα το κάνω. Η πρόεδρος, δεύτερος γύρος ερωτήσεων. Η ε, σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι στην ευτυχή θέση εδώ ότι μιλάω την ίδια γλώσσα με τον υποψήφιο και έτσι μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα, χωρίς τη βοήθεια των διερμηνέων. Είπατε λοιπόν ότι η EBA έχει τις ε, αναγκαίες ε, αρμοδιότητες βάσει του καταστατικού ε, και υπάρχει ήδη μια ροή πληροφοριών μεταξύ εθνικών υποπτικών αρχών και των ευρωπαϊκών αρχών. Πριν, προηγουμένως, ο κύριος Μοντάλβο είπε ότι το πλαίσιο των δραστηριοτήτων σας δυναμητικό έχει ενισχυθεί. Έχει ενισχυθεί πολύ. Θέλω λοιπόν να μας εξηγήσετε γιατί αυτή τη στιγμή η EBA θα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες τραπεζικές αρχές. Ο κύριος Φάρκας. Θα, μι... μιλήσω αγγλικά. Πιστεύω ότι έχουμε θίξει αυτό το ερώτημα και σε προηγούμενα ερωτήματα ε, αυτό το ζήτημα. Ε, η EBA αυτό που έχει ε, σε καινούριο ή περισσότερο σε σχέση με προηγούμενες αρχές είναι νέα μέσα στη διάθεσή της. Οι προηγούμενες αρχές είχαν τη δυνατότητα να προτείνουν και να εκδώσουν συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές. Εκεί όπου διαφέρει η EBA εκτός, ε, ε, ε, παραπάνω δηλαδή, έχει περισσότερες αρμοδιότητες από τις επιτροπές επίπεδου 3, είναι ότι μπορεί να εκδώσει, να συντάξει, να εκδώσει και να εγκριθούν από την Κομισιόν υποχρεωτικοί κανόνες υποχρεωτικοί εφαρμοστικοί κανόνες νομοθετικού περιεχομένου. Αυτό καλύπτει και όλο το πλαίσιο πληρωμών αμοιβών. Επίσης, η EBA θα παρουσιάσει πίνακες αξιολόγησης εντοπισμού κινδύνου, θα εκτελεί ένα αποτελεσματικό ε, ε, ε, μια αποτελεσματική παρακολούθηση και εποπτεία του κολεγίου του σώματος των εποπτικών αρχών που δεν γινόταν στο παρελθόν Επίσης, η EBA μπορεί να αποτανθεί σε μεμονωμένους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ε, και να ζητήσει άμεσα την παροχή στοιχείων εάν η Εθνική Αρμόδια Αρχή δεν τα παράσχει και θα έχει το δικαίωμα να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εάν κάποιος παραβιάζει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ζητήσει την ανάληψη δράσης. Ε, επίσης ε, θα έχει τη δυνατότητα διαιτησίας σε περίπτωση ε, διαφορών και με το παλαιό σύστημα αυτές οι διαφορές που προέκυπταν δεν εμφανίζονταν στην επιφάνεια παρά μόνο την τελευταία στιγμή όταν πια είχε ξεσπάσει μια κρίση σε έναν συγκεκριμένο οργανισμό Εφόσον εμείς τώρα μπορούμε να ε, εφαρμόζουμε την αρχή της διαιτησίας, θα μπορέσουμε να προλαμβάνουμε ε, κρίση σε συγκεκριμένους οργανισμούς ε, και σε διάφορες χώρες. Επίσης έχουμε την εξουσία να απαγορεύσουμε την κυκλοφορία ορισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων ή εφόσον εντοπίσουμε ότι υπάρχει υπερβολικό ρίσκο στην κυκλοφορία ενός επικίνδυνου προϊόντος. Είναι λοιπόν ε, πολύ μεγάλο, δεν μπορώ να σας παρουσιάσω τώρα όλα τα στοιχεία που διαφοροποιούν την EBA από τους προ... τις προηγούμενες αρχές, αλλά αυτές ήταν ορισμένες από τις πολύ σημαντικές νέες ευθύνες και αρμοδιότητες της EBA. Ευχαριστώ. Την επόμενη ερώτηση ο Πίτερ Σκίνερ. Ευχαριστώ, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Από την τελευταία φορά που σας είχαμε δει, είχατε την ευκαιρία να εμπλουτίσετε την πείρα σας και ε, να εμβαθύνετε στα θέματά μας και φαντάζομαι ότι ε, ήταν θετική η εμπειρία σας, αλλά θα ήθελα να κάνω ορισμένες ερωτήσεις και να είμαι και συνεκτικός ε, και ευθύς ε, τελευταίος ε, στον τύπο ε, είπατε ότι είστε μέλος της MTF. Ελπίζω θα μου απαντήσετε γρήγορα σε αυτό, αλλά θα ήθελα να ξέρω αν είσαστε ακόμη σε αυτή την εποπτική αρχή, γιατί αφού το τέλος του 2010 ήσασταν ρυθμιστής, τον Ιανουάριο πώς ήταν δυνατόν να προσληφθείτε κατευθείαν σε μια εταιρεία. Φαντάζομαι ότι θα το εξηγήσετε. Επίσης αυτό που έχω ρωτήσει και σε όλους είναι ότι ε, έχετε 100 άτομα την αρχή που καταρτίζετε θα πρέπει να αξιοποιήσετε στο μέγιστο του σπόρους και πώς θα το επιτύχετε. Πώς δηλαδή θα ε, οργανώσετε τη δουλειά σας. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να απαντήσω διότι έφυγα στην, ε, ε, ε, από τη θέση μου του, στην Ποπτική Ουγγρική Αρχή στα μέσα του 2010 και ε, για αυτούς τους λόγους δεν μπορώ να αναλάβω μία εκτελεστική θέση ε, σε ένα οργανισμό που ποπτεύεται από αυτή την αρχή για λόγους συγκρούσεως συμφερόντων. Οπότε πέρσι τον Νοέμβριο είχα υποβάλει την ε, υποψηφιότητά μου και έχω αναλάβει μία μη εκτελεστική θέση η οποία δηλαδή δεν είναι σε σύγκρουση με ε, τους κανόνες που πρέπει να σεφαστώ είναι εθελοντική εργασία χωρίς οποιαδήποτε εκτελεστική εξουσία ε, και πρέπει να σας πω ότι εντωμεταξύ ήδη έχω υποβάλει την παρέτησή μου, έχω φύγει εφόσον ε, έχω επιτύχει στην υποψηφιότητα και είναι προφανές ότι δεν ε, θα παρέμενα σε μία θέση που θα ήταν σε πλήρη σύγκρουση με αυτήν που επιζητώ το δεύτερο ερώτημα είναι ότι το θέμα σας σχετικά με την EBA είναι ίσως λίγο πολύ αισιόδοξο διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε 100 αλλά θα έχουμε 50 συμβασιούχους ε, υπαλλήλου και θα ε, ε, ελπίζω ότι θα υπάρξουν και 20% που θα διατίθενται ανα πάσα στιγμή πέραν των 50 ατόμων του μονίμου προσωπικού που θα αναλάβει αυτή τη θέση. Από προοπτική μελλοντική η πρόκληση ε, είναι ότι θα μπορέσει να αυξηθεί η αρχή αυτή και να περιλαμβάνει 100 υπαλλήλου σε, σε μία τριετή ε, προοπτική. Υπάρχει θέμα αποτελεσματικότητος και καταρτήσεως προτεραιοτήτων διοικητικών διότι οι εργασίες και τα διάφορα έργα είναι τόσο περίπλοκα ώστε θα υπάρχουν συγκρούσεις ε, μεταξύ των πόρων αυτής της αρχής. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει σωστός προγραμματισμός και συχνή αναθεώρηση των προτεραιοτήτων, να σεβόμαστε τις προτεραιότητες και να τις συνδυάσουμε με πόρους κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε αποτελέσματα και ότι η οργάνωση δεν θα κατακαιρματιστεί υπερβολικά με τις δυνατότητες ε, απολίας ε, των ε, σωστών προτεραιοτήτων και αυτό θα ήταν μία από τις βασικές μου ε, ευθύνες να εξασφαλίσω ότι οι πόροι που διαθέτουμε θα χρησιμοποιηθούν με τον καταλληλότερο και τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Ευχαριστώ. Γουλφ Κλίντ, αλλά φαντάζομαι ότι εγώ θα μιλήσω στο σημείο αυτό. Θα ήθελα να επανέλθω σε ένα ερώτημα το οποίο έθεσε η Σιλβί Γκουλάρ και που είχε να κάνει με τη διαχείριση των κρίσεων, με το καθεστώς διαχείρισης των κρίσεων. Το ότι το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας για το ευρώ και άλλοι παράγοντες ουσιαστικά έχουν ε, αναλάβει, έχουν σπρώξει κάποιες αρμοδιότητες πίσω στα κράτη-μέλη, όσον αφορά για παράδειγμα την ε, επανακεφαλαιοποίηση τραπεζών κτλ αλλά άκουσα προσεκτικά την απάντησή σας και σας άκουσα να λέτε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη επικοινωνία και μεγαλύτερη έκθεση στο νέο καθεστώς τεστ αντοχής για τις τράπεζες, ιδίως όσον αφορά τα ομόλογα. Και Αναρωτιέμαι αν όντως θέλετε να πετύχετε ένα υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας και αν θέλετε να πετύχετε και ένα καλύτερο συσχετισμό όχι μόνο αυτό που υπάρχει ανάμεσα στις τράπεζες και το δημόσιο χρέος αλλά και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ τραπεζικών προϊόντων από τη μία τράπεζα στην άλλη αυτή η αλληλοέκθεση που υπάρχει μεταξύ τραπεζών είναι πάρα πολύ σημαντική ως προς την αντιμετώπιση της κρίσης. Όταν καλούμεθα να αποφασίσουμε πώς πρέπει να γίνει η αναδιάρθρωση του κεφαλαίου μιας τράπεζας, ξέρω ότι δεν αποτελεί αυτό άμεση αρμοδιότητα της EBA, αλλά θα ήθελα τη δική σας προσωπική τοποθέτηση. Απάντηση, σας ευχαριστώ. Επανερχόμενος ε, στα σχόλιά σας για το καθεστώς διαχείρισης των κρίσεων, θα έλεγα ότι οι πρόσφατες εξελίξεις που έχουμε, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, θα οδηγήσουν σε μία λύση που θα είναι ουσιαστικά ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την διαχείριση των κρίσεων. Ως προς αυτό λοιπόν συμφωνώ με τις δικές σας προσπάθειες και τη δική σας τοποθέτηση εν γέννη. Όντως είναι σαφές ότι οι εθνικές λύσεις που προτάθηκαν δεν αρκούσαν για την αντιμετώπιση της κρίσης και ας μην ξεχνάμε ότι η διαχείριση των κρίσεων δεν έχει να κάνει μόνο με την διάσωση τραπεζών που έχουν πτωχεύσει. Υπάρχουν πολλά άλλα βήματα τα οποία πρέπει να καλύψει κανείς προτού φτάσει εκεί. Επομένως μια ευρωπαϊκή προσέγγιση θα πρέπει να υπάρχει και θα πρέπει να εγκρίνεται σε έναν ε, πρώιμο σημείο, χρονικό σημείο, πρωτού φτάσουμε δηλαδή στην κρίση, προτού χρειαστούν δηλαδή τα χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογουμένου για να διασωθεί μια τράπεζα. Όσον αφορά τη διαφάνεια τώρα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η οικονομική κρίση κατέδειξε, και ιδίως η πτώση των Lehman Brothers, ότι ε, μία από τις σημαντικότερες ε, δυσκολίες όλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος και ένας από τους σημαντικότερους λόγους ε, της ε, κατάρρευσης ε, του συστήματος ήταν ότι, τα, ότι οι ίδιοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δεν γνωρίζανε σε ποιο βαθμό είχαν εκτεθεί σε σχέση με άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι ε, φάνηκε κατά αυτόν τον τρόπο τόσο έντονα η έλλειψη διαφάνειας στην αλληλοσύνδεση αυτή που υπάρχει μεταξύ τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Ακόμα και οι ρυθμιστικές αρχές δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν ακριβώς πώς το δικό τους εποπτικό σύστημα ή το δικό τους τραπεζικό σύστημα είχε εκτεθεί ως προς ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή μια τράπεζα. Το να αυξήσουμε λοιπόν τη διαφάνεια όσον αφορά την έκθεση, όσον αφορά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία όσον αφορά την ε, κεφαλιακή σύνθεση των τραπεζών, όσον αφορά την έκθεσή τους σε άλλους παράγοντες στο τραπεζικό τομέα. Η διαφάνεια λοιπόν αυτή θα μας οδηγήσει σιγά σιγά σε ένα καλύτερο κλίμα αμοιβέ εμπιστοσύνη των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα θα έχουν μάλλον μια πιο ξεκάθαρη εικόνα οι εθνικές εποπτικές αρχές στην αξιολόγηση που καλούνται να κάνουν κάθε φορά που ε, εμφανίζεται σιγά σιγά μια κρίση, είτε πρόκειται για μια οικονομική κρίση χώρας, είτε πρόκειται για συγκεκριμένη κρίση που αφορά συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Σα Σας ευχαριστούμε πολύ. Γιώργη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Φάρκας, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Τρεις πολύ σύντομες ερωτήσεις όσον αφορά το συστημικό κίνδυνο καταρχάς. Και έπειτα στη συνέχεια, οι πόροι προχρηματοδότησης για ορισμένες επενδύσεις και έπειτα το ζήτημα του δημοσίου χρέους και των κεφαλαίων που απαιτούνται ως προς αυτό. Για το πρώτο όμως ζήτημα, το ζητήσαμε πάρα πολύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συστημικό κίνδυνο δηλαδή, και θελήσαμε να δούμε ποια θα είναι τα κριτήρια αυτά, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τους τη διάσταση του κινδύνου και πώς θα μπορούσαμε να είχαμε και ένα καθεστώς τεστ αντοχής. Τα στοιχεία αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά προκειμένου να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα. Χρειαζόμαστε προφανώς κανόνες οι οποίοι θα υλοποιούνται και θα εφαρμόζονται από όλου και θα πρέπει να συνοδεύονται από τον κατάλληλο μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το ακόλουθο. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που θα χρησιμοποιεί καταλόγους, θα πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα αντιμετώπισης κρίσεων, δηλαδή ένα σύστημα το οποίο να είναι κομμένο και ραμμένο στις ευρωπαϊκές ανάγκες, να αντιμετωπίζει τις ιδιοσυγκρασίες του ευρωπαϊκού συστήματος. Και έπειτα, Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ταμείο εγγύηση καταθέσεων το οποίο να συνδέεται με τα εθνικά αντίστοιχα ταμεία και ένα ξεχωριστό επιταταμείο για την επίλυση των κρίσεων. Μιλάω πάντα για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα ταμείο μάλιστα το οποίο να έχει ένα ανοιχτό πεδίο εφαρμογής. Είναι πολύ δύσκολο να επιλύσει κανείς μια παγκόσμια διασυνοριακή κρίση με τόσα πολλά χρηματοπιστωτικά, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς κάθε φορά που μιλάμε για διασυνοριακές συναλλαγές. Το σύστημα το οποίο έχει εγκριθεί αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών κρίσεων έχει λάβει υπόψη του τις χώρες που έχουν ένα σημαντικό πρόβλημα δημοσίου χρέους. Αν λάβουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες λοιπόν του χρέους αυτού, Θα πρέπει να εξετάσουμε στην περίπτωση αυτή τα αποθεματικά τα οποία θα πρέπει να έχουμε διαθέσιμα και ουσιαστικά θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διασυνδέσουμε το μηχανισμό αυτό αντιμετώπισης του δημοσίου χρέους, κρίσης δηλαδή που συνδέεται με το δημόσιο χρέος, με το τραπεζικό σύστημα το οποίο θέλουμε να έχουμε στο μέλλον στην Ευρώπη. Μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα αυτό. Um, I'm not sure I δεν είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα ακριβώς τη συγκεκριμένη ερώτησή σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και αν δεν σας καλύψω θα ανταπαντήσω. Με το θέμα ε, της εγγύησης των καταθέσεων και το αντίστοιχο ψήφισμα ε, αυτό συνάδει με αυτά που είπα προηγουμένως. Η μακροπρόθεσμη λύση με τον μεγάλο αριθμό των ε, διατραπεζικών ε, συναλλαγών που γίνεται στην Ευρώπη, πολλές τράπεζες που λειτουργούν διασυνοριακά, η λύση του προβλήματος αυτού θα ε, παρουσιαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να βρεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα διότι ε, θα πρέπει να ληφθούν ε, δύσκολες αποφάσεις, δηλαδή πώς ε, αυτό το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων θα χρηματοδοτηθεί, θα, θα είναι μέσα στο πλαίσιο της σύγχρηματοδότησης, τι πόρους θα έχει και τι αποφάσεις θα ληφθούν για τη χρήση, χρήση αυτού του ταμείου. Είναι ένα ε, ζήτημα με σοβαρές πολιτικές πτυχές. Οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για τη λειτουργία αυτού του ταμείου είναι πολιτικές. Όσον αφορά τώρα το εθνικό χρέος, τα εθνικά χρέη, και, και τις κεφαλογικές ανάγκες Νομίζω ότι τα δύο αυτά συνδέονται. Η, τα, εθνικά το, κυρίαρχο χρέος, το sovereign debt ε, ε, συνδέεται με τις κεφαλαιοχικές ανάγκες. Το ψήφισμα, το Συμβούλιο και, και το Κοινοβούλιο στο το ψήφισμα λέει ότι θα πρέπει να βρηθούν κριτήρια για την επισήμανση συστημικού ρίσκου τα οποία θα πρέπει να εποπτεύει το ΙΜΠΑ και να προτείνει συγκεκριμένο μηχανισμό λύσεων. Τι, πώς νομίζετε, τι νομίζετε ότι καλύπτει αυτή η ενισχυμένη εξουσία της ΙΜΠΑ για την ανάλυση συστημικών ρίσκων και την εξέβρεση λύσεων ο κύριος Φάρκας. Εγώ νομίζω ότι η επισήμανση αυτών των κινδύνων, αυτών των συστημικών προβλημάτων που προκύπτουν από ένα συγκεκριμένο οργανισμό μπορούν να προέλθουν από διαφορετικές πηγές. Πρώτον, η επισήμανση αυτή του συστημικού κινδύνου μπορεί να προέλθει από την ECRB, μπορεί να προέλθει από μια εθνική αρχή ή από τον Ευρωπαϊκό Φορέα Ανάλυση Συστημικών Ρίσκων λοιπόν και να υποβληθεί στην EBA ε, μπορεί να έρθουν λοιπόν από διάφορους, διάφορες πηγές ε, αυτή η ένδειξη και η ίδια η EBA μπορεί όταν θα εκτελεί ένα, τραπεζικό, ένα τεστ τραπεζικής αντοχής να επισημάνει ε, ένα συστημικό κίνδυνο και να σηκώσει την κόκκινη σημαία να εκπέμψει σήμα κινδύνου. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε τότε είναι να το ε, φέρουμε εις γνώση του, ε, του Διοικητικού Συμβουλίου Εποπτικών Αρχών ε, και να αποφασίσει και να αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως EBA. Οπωσδήποτε πρέπει να κοινοποιήσουμε άμεσα τις εθνικές αρχές για αυτό τον κίνδυνο που επισημάναμε. Το ESRB επίσης, αυτό τον Ευρωπαϊκό Φορέα ε, Συστημικών Κινδύνων πρέπει επίσης να γνωσ... κοινοποιήσουμε ε, και το κολέγιο, αυτό το, ε, το σώμα ρυθμιστικών αρχών πρέπει να λάβει γνώση και Εάν η ενδεχόμενη κρίση είναι πάρα πολύ σοβαρή, η EBA μπορεί να ξεκινήσει ε, την, ε, να ξεκινήσει την διαδικασία ε, κατεπίγουσας ε, δράσης μαζί με το Συμβούλιο. Εάν, εάν λοιπόν αναγνωριστεί ότι είναι κατεπίγουσα η κατάσταση αυτή, τότε η EBA θα λάβει μέτρα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, Ελίσσα. Ευχαριστώ για όλες αυτές τις προφορίες και τις ιδέες που μας παρουσιάσετε. Θέλω να επανέλθω στην, ε, στο πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων. Ε, έχοντας υπόψη και αυτό που είπε ένας άλλος συνάδελφος προηγουμένως, το Κοινοβούλιο σε μία έκθεση πρωτοβουλίας ξεκάθαρα απέτησε τη δημιουργία ενός κοινού ταμείου έτσι ώστε να μην φορτωθείτε εσείς προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν μέσα στο τραπεζικό σύστημα. Εν τω μεταξύ βλέπουμε πάρα πολλά μηνύματα, πολλά σημάδια ε, από πλευράς Συμβουλίου ε, το Μάρτιο τώρα πρόσφατα αλλά και πριν ότι δημιουργείται μια εθνική προσέγγιση προς αυτό. Τι μπορεί λοιπόν η EBA να κάνει για να μην χαθεί αυτή η κίνηση δημιουργίας ενός πραγματικά ευρωπαϊκού πλαισίου να λυθεί αυτή η κατάσταση. Δεύτερη ερώτηση. Εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία στην αγορά χρεογράφων και αυτό πιστεύω ότι αξιολογήθηκε πολύ σωστά διότι εργαστήκατε χρόνια στο τραπεζικό τομέα και καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Πιστεύετε ότι αυτό βοηθάει ή όχι, διότι ε, οι περισσότεροι κίνδυνοι Στι τράπεζε προέρχονται από άλλε πηγές και δεν είναι μόνο εσωτερική κίνδυνη που δημιουργήθηκαν στην τράπεζα. Νομίζω ότι συμφωνώ μαζί σας με την παρατήρηση που κάνατε ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική όρεξη η, η πρόθεση των ε, εθνικών αρχών για να, να συμφωνήσουν σε ένα κοινό ταμείο μειώνεται. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα του και τις γνώσεις του για να διατυπώσει προτάσεις για να μπορέσει αυτό, αυτή η διαδικασία να επανέλθει στο προσκήνιο. Βεβαίως ε, εδώ μιλάμε για την ε, τραπεζική αρχή. Ε, οπότε πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θα είναι ένας βασικός παίκτης για να παραμείνουν τα θέματα στη συζήτηση, στο προσκήνιο με τεχνικά και σωστά επιχειρήματα και δεν πρέπει να σταματήσει ε, λόγω μίας επιβραδύνσεως της διαδικασίας εάν οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να προχωρήσει. Όσον αφορά τις αγορές Πιστεύω ότι χωρίς να γνωρίζουμε την αγορά των ε, χρεογράφων είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε τον τομέα των τραπεζών διότι τα τελευταία 20 χρόνια έχει υπάρξει μεγάλη ροή η μεγάλη διαδικασία ε, εξελίξεως των χρεογράφων πολύ κίνδυνοι διατυπώνεται μέσω χρεογράφων και πολλά από αυτά απορρέουν από τους ισολογισμούς των τραπεζών και διαμορφώνουν χρεόγραφα και τα νάπαλιν. Ε, τα χρεόγραφα περιλαμβάνονται στους ισολογισμούς των τραπεζών. Οπότε σε αυτή σε αυτό το τομέα η αρχή θα μπορούσε να βοηθήσει και η συνεργασία μεταξύ του υπευθύνου για τα χρεόγραφα και του υπεύθυνη αρχής για τις ε, τράπεζες ε, θα μπορέσει επίσης να βοηθήσει διότι θα καταργηθούν τα στεγανά και θα μπορεί ο καθένας να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συστημιατικών προβλημάτων. Νομίζω ότι τώρα έχουμε καλύψει το χρόνο μας και ο Γκέφχαρτ είναι ο τελευταίος που έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομος, αλλά έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση, Βασιλεία 3 πώς εσείς αντιμετωπίζετε την εφαρμογή της Βασιλείας 3 ή στο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρχει ισότιμο παιχνίδι στην Ευρώπη. Δηλαδή εάν άλλες χώρες εκτός Ευρώπης δεν εφαρμόσουν τη Βασιλεία 3 πώς θα πρέπει εμείς να συμπεριφερθούμε στην Ευρώπη. Δεύτερον, αν σας επιβεβαιώσει το Κοινοβούλιο πώς εσείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να διατυπώσετε κατευθυντήριες γραμμές προς την τραπεζική αρχή και όπως όπως ε, είπε και ο Πίτερ Σκίνερ ε, ε, είδα το βιογραφικό σας αλλά βρέπω ένα κενό μεταξύ 95 και 97 τι κάνατε την περίοδο 95 με 97 Σας ευχαριστώ θα απαντήσω στο πρώτο σας ερώτημα που έχει να κάνει με την παγκόσμια εφαρμογή της Βασιλείας 3. Η θέση της Ευρώπης και των οργάνων που έχουν ως ρόλο τους να εφαρμόσουν τη Βασιλεία 3 πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Αν η Συμφωνία Βασιλεία 3 είναι διεθνής συμφωνία με την οποία έχουν συμφωνήσει τελικά όλα τα συμβαλώμενα μέρη σε όλες τις περιοχές του κόσμου, τότε ξέρουμε ότι χρειάστηκε να δοθούν σημαντικές μάχες για να καταλήξουμε στη συμφωνία αυτή, αλλά καταλήξαμε συμφωνία αυτή με όλο το χρονοδιάγραμμα το οποίο προβλέπεται για την εφαρμογή της, τότε η Ευρώπη θα πρέπει να επιμείνει για την υλοποίηση, για την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής από όλα τα συμβαλόμενα μέρη, σε όλες τις περιοχές. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα σαφές μήνυμα το οποίο θα πρέπει να στείλει ως προς τη Βασιλεία Τρία η Ευρώπη στο σύνολό της. Το δεύτερο ερώτημά σας είχε να κάνει με την αποστολή που θα έχουν οι εργαζόμενοι στην EBA το βασικό μήνυμα εδώ είναι ότι η αρχή αυτή έχει πολύ υψηλές προσδοκίες, έχει πολλά ενδιαφέροντα καθήκοντα, μια ευρή εντολή και νομίζω ότι θα πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε αποτελέσματα, ότι δηλαδή η δημιουργία της CBA ήταν όντως ένα πολύ θετικό βήμα και θα ήθελα να κινητοποιήσω όλους τους συναδέλφους μου προκειμένου να εργαστούν με τα υψηλότερα δυνατά επαγγελματικά κριτήρια, να, έχουν, να δείξουν ένα απόλυτο βαθμό ακαιρεότητας και ανεξαρτησίας στην καθημερινή τους εργασία και από την άλλη όμως πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να είναι ένας ενδιαφέρον χώρος όπου μπορεί κανείς να εργάζεται με ενθουσιασμό. υπάρχει δηλαδή το κατάλληλο επαγγελματικό περιβάλλον. Τώρα, αναφερθήκατε στο βιογραφικό μου και στο κενό το οποίο εμφανίζεται μεταξύ 95 και 97. Δεν έχω μελετήσει πολύ καλά το σημείο αυτό. Ήμουν πάντω καθηγητή μέχρι να πάω στην Κεντρική Τράπεζα τη Ουγγαρία. Εργαζόμουν πλήρω ω καθηγητή ε, χρηματοπιστωτικών οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της ε, Βουδαπέστης. Σα Σας ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώθηκε κατά αυτόν τον τρόπο γύρω των ερωτήσεων. Έχετε προφανώς τη δυνατότητα να ξαναπάρετε το λόγο αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, αν θέλετε να συνοψίσετε λίγο την παρέμβασή σας. Έχετε ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος. Δεν έχουμε σεβαστεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Ολοκληρώνω λοιπόν λέγοντας, ε, μάλλον ευχαριστώντας σας για τη δυνατότητα που μου δώσατε να έχω την πολύ αυτή ενδιαφέρουσα ουσιώδη ανταλλαγή απόψε, να ακούσω τις ουσιώδεις ερωτήσεις σας. Προσβλέπω στην υποστήριξή σας και εφόσον ε, με επιβεβαιώσετε στη θέση αυτή, προφανώς θα επιστρέψω στην Επιτροπή σας και θα σας ενημερώσω για τις επιτυχίες, και επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Σας ευχαριστώ πολύ. So, σα ευχαριστούμε. Λοιπόν, πώς έχει τώρα η διαδικασία. Θα συνεδριάσουμε σύντομα και κλεισμένων των θυρών. Επομένως όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να αποχωρήσετε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να καταναλώσουμε πάρα πολύ χρόνο. Πάρα πολλά ζητήματα καλύψαμε ήδη χθες.